Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε γιατί συμφωνήσαμε χθε να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε στην ώρα μας όσο γίνεται. Εν πάση περιπτώσει. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε και να καλωσορίσω θερμότατα τον Επίτροπο και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φυσικά και τα κρατήρα, τους καλεσμένους μας, τους ευρωβουλευτές. Έχουμε και καλεσ... καλεσμένος κυρία Σράιερ. Καλώς ήρθατε. Ήρθατε σε μια πολύ καλή στιγμή για να ακούσετε και την ομιλία του Επιτρόπου Χόγκαν με θέμα το οικολογικό σχεδιασμό των στρατηγικών σχεδίων της κοινή γεωρικής πολιτικής. Ένα θέμα που εγείρει πολλά ερωτήματα. Πώς θέλουμε να συνδυάσουμε αυτά τα οικολογικά προγράμματα και τα μέτρα του δεύτερου πυλώνα, για παράδειγμα. Τι ακριβώς ε, είναι υποχρεωτικό. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τη διπλή χρηματοδότηση. Και Επίσης, ε, η σημερινή ανταλλαγή απόψεων έγινε πρωτοβουλία του Επιτρόπου και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερως γι' αυτό. Γιατί θέλουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τους ευρωβουλευτές αλλά και τους καλεσμένους ε, που πολύ συχνά παρακολουθούν τις εργασίες μας. Αυτά ευχαριστώ και ο λόγος στον Επίτροπο Χόγκαν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, κυρίε και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω πάλι στην Επιτροπή σας όπου εργάζεστε σκληρά για να υπάρξει μια πρόοδος για την ΚΑΠ μετά το 2020. Ειδικά το τι θα κάνει η μελλοντική ΚΑΠ σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Και δικαίω. Την προηγούμενη εβδομάδα αρκετοί άνθρωποι εδώ πέρα είδαν και άκουσαν γύρω στους 12.000 φοιτητέ που διαδήλωσαν και ζητούσαν να γίνει κάτι για την κλιματική αλλαγή. Την ίδια στιγμή ακριβώς που έχουμε νέες προειδοποιήσεις για την βιώσιμη και μη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων σε ένα επιστημονικό περιοδικό και ένα άλλο περιοδικό το οποίο έλεγε ότι η γεωργία είναι το νέο κάπνισμα. Δηλαδή η κοινωνία αναμένει μεγάλες άλλαγες στην βιωσιμότητα της γεωργίας ε, και στα ζητήματα περιβάλλοντος. Και ελπίζουμε βεβαίως αυτά να τα υλοποιήσει η ΚΑΠ. Δεν πρέπει επίσης να χάνουμε... Να ξεχνάμε την σκοπιά του προϋπολογισμού, όπου προωθούνται οι συζητήσεις, αλλά οπωσδήποτε θα προσπαθήσω να υπερασπιστώ τον προϋπολογισμό της Γεωργίας. Πιστεύω λοιπόν ότι η πρόταση της Κομισιόν θα αλλάξει τα πράγματα όσον αφορά την καλύτερη απόδοση και τα καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα του κλίματος, του περιβάλλοντος και της αηφορίας. Οι υπηρεσίες μου έχουν συντάξει ένα νέο έγγραφο, το οποίο σας μοίρασαν σήμερα για να ξεκαθαρίσουν διάφορα ζητήματα και βεβαίως ε, εξηγεί και κάποια ζητήματα που αναφέρονται στις ε, τροπολογίες. Λέει πώς ακριβώς θα έχει σοβαρότερα ωφέλη η ΚΑΠ και ταυτόχρονα θα καταστήσει πιο καλή την προστασία του περιβάλλοντος. Ε, σας έχουμε δώσει αυτό το έγγραφο και γι' αυτό τον λόγο δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα να τονίσω ορισμένα σημεία. Πρώτα απ' όλα, να σας πενθυμίσω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αφορούν την κλιματική αλλαγή, την αντιμετώπιση και την προσαρμογή, δηλαδή το νερό, ποιότητα και ποσότητα, τον αέρα και το χώμα, την βιοπικιλότητα και τα τοπία. Αλλά επίσης είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον γενικότερο στόχο μας για να διασφαλίσουμε την διατροφική ασφάλεια για τους ανθρώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την δυνατότητα βεβαίως των αγροτών να μπορούν να ζήσουν από τη δουλειά τους. Οπότε, η προστασία του εδάφου ή η προστασία της βιοπικιλότητας, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά ζητήματα. Αφορούν απευθεία και άμεσα την γεωργία και την ε, ικανότητά μας να προστατεύσουμε τη δυνατότητα παραγωγής τροφίμων και στο μέλλον. Οπότε βλέπετε εδώ πέρα συνοπτικά τρει στόχου που προτείνει η Κομισιόν. Βεβαίω ε, συζητάμε ακόμα τις ε, διατυπώσεις και τις λεπτομέρειες, αλλά ελπίζω να συμφωνήσετε στις αρχές. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής, των φυσικών πόρων και της βίοποικιλότητας. Γιατί χωρίς αυτά δεν θα έχουμε βιώσιμα αγροκτήματα και άρα αγρότες. Εάν συμφωνούμε σε αυτό το βασικό, τότε έχουμε κάνει κάποια πρόοδο. Το κοινό, η κοινή γνώμη ζητά ακριβώς να κάνουμε κάτι για αυτούς τους στόχους. Το διάγραμμα αυτό μας δείχνει απλά το πώς ε, θα προσπαθήσει να επιτύχει τους στόχους η ΚΑΠ σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα. Μας υπενθυμίζει εδώ πέρα πως ε, οι βελτιώσεις δεν αφορούν μονάχα τα αποτελέσματα του νέου μοντέλου, αλλά και τις βελτιώσεις της ήδη φυστάμενης για την νέα εργαλειοθήκη, αλλά και την καινοτομία και την ψηφιοποίηση. Όσον αφορά τα αποτελέσματα και το νέο αυτό μοντέλο, αυτό από μόνο του αξίζει μια πλήρη συζήτηση, αλλά για την σημερινή συζήτηση θα ήθελα να τονίσω ότι είναι σημαντικό ότι σύμφωνα με το νέο μοντέλο τα κράτη-μέλη θα προσαρμόσουν μια ευρύτατη στρατηγική που θα περιλαμβάνει και τους δύο πυλώνες της ε, ΚΑΠ, μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με την σημερινή κατακαιρματισμή προσέγγιση. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σε μια ανάλυση των ισχυρών σημείων, των ε, ασθενέστερων σημείων και των ευκαιριών και των κινδύνων που έχουμε με βάση τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας. Και σκοπεύουμε ακριβώς να βασιστούμε σε στόχους που έχουμε ήδη και χρησιμοποιούμε δείκτες, ε, οι τιμές των οποίων θα καθοριστούν από το τι κάνουν τα κράτη-μέλη αντί για εξωτερικούς παράγοντες. Οπότε θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι αναμένουμε μια στόχο θυσία η οποία θα είναι υπεύθυνη και φιλόδοξη από τα κράτη-μέλη είναι δική του ευθύνη, αλλά βεβαίω και η Κομισιόν θα αξιολογήσει τα όσα προτείνουν. Αλλά ουσιαστικά ακούω κόσμο να ζητάει περισσότερη ευελιξία για του αγρότε και η συζήτηση για το Omnibus ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχετε μια αίσθηση ότι το υφιστάμενο σύστημα με όλα του τα ελαττώματα είναι ένα καλό συμβασμό. αλλά σα διαβεβαιώ ότι το ακριβώ το σκεπτικό, το να δώσουμε περισσότερα ευελιξία στου αγρότες, είναι αυτό το οποίο οδηγεί σε περισσότερη επικουρικότητα. Έχουμε λοιπόν μια ρητή αναφορά στην σχέση τη ΚΑΠ με το κλίμα και θα έχουμε έτσι μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τη πολιτική για να διασφαλίσουμε ότι θα έχει μέλλον η γεωργία. Οπότε η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Όταν ένα κράτο μέλο λοιπόν συντάσσει το στρατηγικό του σχέδιο θα λαμβάνει υπόψη την ανάλυση που αλλά γίνεται από τις ε, διάφορες οδηγίες όπως η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα κτλ. Και τότε θα παρουσιάζει ξεκάθαρα την συνεισφορά της γεωργίας για την επίτευξη αυτών των στόχων με βάση την νομοθεσία αυτή. Πρόκειται λοιπόν για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Κατόπιν περνάμε στην αιρεσιμότητα, κάτι το πολύ σημαντικό. Γνωρίζω ότι κάποιες ίσως από τις προτάσεις της Κομισιόν θεωρούνται υπερβολικές όσον αφορά το περιβάλλον, αλλού θεωρείται ότι δεν κάνουμε αρκετά. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί η σωστή ισορροπία. Η αιρεσιμότητα θα αποτελέσει μια βάση των όσων θα επιτύχει για το περιβάλλον και το κλίμα η ΚΑΠ. Ε, Ένα θεμέλιος λίθος θα έλεγα. Οπότε πρέπει να είναι στιβάρος ως ε, θεμέλιος λήθος, αλλά προτείνουμε ταυτόχρονα να επιτύχουμε μια ισορροπία, Παράδειγμα του χάρη για τους υγροτόπους ε, και τις εκτάσεις με τύρφη που συλλέγουν ε, διοξίδιο του άνθρακα. Έχουμε κάποιους περιορισμούς όσον αφορά την χρήση ζανιοκτώνων που μπορούν να ενταχθούν στην αιρεσιμότητα και έχουμε ακριβώς ε, την ψηφιοποίηση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στον τομέα αυτών για την χρήση των διαφόρων λιπασμάτων χωρίς να έχουμε περίπλοκες υποχρέωσει για τους αγρότες. Το ίδιο και για τις περιοχές όπου έχουμε προτείνει να υπάρξει μια προσαρμογή της λεγόμενης πολλαπλής συμμόρφωσης, παραδείγματος χάρη. Ε, η πρόταση για να περάσουμε στην άμυψη σπορά από το προηγούμενο σύστημα νομίζω ανταποκρίνεται στις ανησυχίες οποίες εκφράσατε και εσείς. Ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη θα έχουν επαρκή ευελιξία για να εφαρμόσουν ε, τις απαιτήσει ε, της αιρεσιμότητας ανάλογα με την κατάσταση του καθενός. Δεν θα έχουμε πλέον τους πολύ περιγραφικούς κανόνες του πρασινίσματος που είχαν ατελείωτους ε, καταλόγους. Ανταυτού θα τα εφαρμόζουμε με βάση στοιχεία και ένα συνεπές σχέδιο για την ΚΑΠ για να έχουμε περισσότερους αγρότες οι οποίοι θα εμπλακούν έτσι ώστε ο αγροτικός κόσμος να μπορεί να ανταποκριθεί στις ε, προκλήσεις. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα έχουμε μεγαλύτερη συγκρισιμότητα και διαφάνεια μεταξύ των κρατών μελών και ίσως όρους ανταγωνισμού. Και πραγματικά πιστεύω ότι η πρόταση αυτή για την αριθμότητα είναι αναλογική και ισορροπημένη σε σχέση με τους συνολικούς μας στόχους. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα στοιχεία της ε, ΚΑΠ τα οποία βασίζονται στα θεμέλια που έχουμε ήδη θέσει. Μεταξύ αυτών βεβαίω είναι και τα οικολογικά συστήματα, τα οποία είναι κάτι το καινούριο πραγματικά στην εργαλειοθήκη μας για το περιβάλλον. Ναι, πράγματι, έχουν κάποια κοινά στοιχεία με τις πληρωμές για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα στον πυλώνα 2, αλλά δεν είναι το ίδιο. Το επεξηγηματικό έγγραφο το οποίο έχετε παρουσιάζει τις διαφορές, αλλά θέλω να τονίσω εδώ πέρα τρία πράγματα. Πρώτα, πληρώνονται πλήρως από τον προπολογισμό του πυλώνου 1, οπότε απαιτούν μηδενική συγχρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, ουσιαστικά λειτουργούν μέσω ετήσιων δεσμεύσεων και όχι πολυετών. Έτσι μπορούν να υποστηριχθούν αγρότες οι οποίοι θέλουν να δοκιμάσουν κάτι για ένα-δύο χρόνια και μετά μπορούν να αλλάξουν ε, κατεύθυνση χωρίς να χάσουν το εισόδημά τους και χωρίς να δεσμεύονται για μια μακροχρόνια περίοδο. Τα κράτη-μέλη θα έχουν ευελιξία όσον αφορά την μορφή των ε, πληρωμών, έτσι θα μπορούν να προσφέρουν κίνητρα στους αγρότες. Υπό τον όρο και Βεβαίω ότι θα σέβονται του σχετικού κανόνε του πράσινου κουτιού του ΠΟΕ. Και βεβαίω τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν και το περιεχόμενο των οικολογικών αυτών έργων σύμφωνα με την κατάστασή του. Οπότε θεωρώ ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα σε πολλού τομεί. Και θα υπάρξει μια ουσιαστική αύξηση στην έκταση που θα καλύπτεται από τα περιβαλλοντικά μέτρα σε σχέση με το τι γίνεται τώρα στον πυλώνα 2. Θα έχουμε λοιπόν μια αποτελεσματική χρήση των εργαλείων αυτών που θα συνδυάζει ακριβώς τα οικονομικά ωφέλη με τα περιβαλλοντικά. Έρχομαι τώρα στον πυλώνα 2. Όπως αντιλαμβάνομαι μέχρι τώρα τις συζητήσεις, λίγοι λένε ότι έχει μεγάλα κενά ε, ο προτινόμενος πυλώνας 2. Ανταυτού εστιάζονται σε διάφορες μεμονωμένες πτυχές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον πυλώνα 2. Κάποιοι προτείνουν να βάλουμε περισσότερες λεπτομέρειες στους κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παραδείγματος χάρη όσον αφορά το τι είδου πληρωμές μπορούν να στηρίξουν τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Εγώ όμως είμαι εναντίον, καθώ δεν θέλω να γίνει πιο πολύπλοκη πολιτική. Εντό του προτινόμενου νέου μοντέλου προσπαθούμε να αποφύγουμε καταστάσει όπου οι πανευρωπαϊκοί κανόνε δεν θα τα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα στο πεδίο που διαφέρει από κράτο μέλο σε κράτο μέλο. Και βεβαίω θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου, όταν μιλάμε για τον πυλώνα 2, ότι οι στραματικές πληρωμές δεν είναι πάντα όλη η αλήθεια. Χρειάζεται εκπαίδευση, συμβουλές, ε, καινοτομία, αγρότες και λοιποί να συνεργάζονται και μόνο με τη χρήση όλων αυτών των εργαλείων η ΚΑΠ θα επιτύχει τα όσα μπορεί. Οπότε μιλάμε για τα οικολογικά αυτά σχέδια τα οποία είναι υποχρεωτικά για τα κράτη-μέλη, εθελοντικά για τους αγρότες, με κάποια κίνητρα αντί για ε, υποχρεωτικούς κανόνες όπως έχουμε σήμερα στο πρασίνισμα. Να σας δώσω λοιπόν κάποια παραδείγματα. Το πρώτο φορά την βιοπικιλότητα. Ε, εδώ πέρα λοιπόν έχουμε πληροφορίε, ε, δεν είναι περιπλοκότητα. Είναι από το έγγραφο το οποίο έχετε μπροστά σα. Δεν θα μπω λοιπόν στι λεπτομέρειε, αλλά μα δείχνει το τι μπορούμε να κάνουμε σε ένα υποθετικό παράδειγμα ενό ε, κράτου μέλου για την εφαρμογή τη βιοπικιλότητα. Μα δείχνει πώ η ευελιξία την οποία προσφέρουμε στα κράτη-μέλη θα λειτουργήσει. Έχουμε για την κλιματική αλλαγή επίσης την προσαρμογή και την αντιμετώπιση. Τα περισσότερα σχόλια σήμερα αφορούσαν το περιβάλλον και το κλίμα. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για την απλοποίηση. Προσπάθησα με την δευτερογενή νομοθεσία να φέρουμε κάποιε αλλαγέ στην πολιτική και θέλω να τονίσω ότι αυτό θα συνεχιστεί με την βοήθειά σας για να ωφεληθούν οι αγρότες. Το να έχουμε λιγότερους ε, και λιγότερο περίπλοκους ε, κανόνες πραγματικά θα βοηθήσει τους αγρότες να ανταποκριθούν ανάλογα με την κατάσταση του καθενός και να μπορούν να παράγουν και να ε, βγάλουν το βιό τους οι άνθρωποι. Όπως ήδη έχω υπογραμμίσει, υπάρχουν κάποια νέα είδη στήριξη, ε, τα οποία θα βοηθήσουν τους ε, αγρότες να έχουν τις στήριξη που χρειάζονται και να ασκήσουμε αποτελεσματική πολιτική. Στη συνολική αυτή προσέγγιση έχουμε διαχείριση, ελέγχους και κυρώσεις που θα είναι ελαφρύτερες, πολύ ελαφρύτερα λεπτά Και θα χρησιμοποιούμε και την πληροφορική, τηλεπισκόπηση και τα σχετικά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, παράδειγμα τους χάρη, για να περάσουμε στην άμυψη σπορά στο μελλοντικό σύστημα. Οι κανόνες σήμερα είναι πάρα πολύ περιγραφικοί και λεπτομερείς όπως βλέπετε. Περιγράφουν τους ορισμούς ε, των φυτών ε, ε, που φυτεύει κανείς, ε, την έκταση και τα σχετικά. Ενώ με την σφορά επαφίεται στο κράτος μέλος να ορίσει κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, καταλήγοντας, η νέα πράσινη αρχιτεκτονική κατά την απόψή μου είναι μια μεγάλη βελτίωση για τους αγρότες και για το περιβάλλον. Δίνει περισσότερες ευκαιρίες για να πληρωθούν οι αγρότες οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν δημόσια αγαθά, απλοποιεί τα περιβαλλοντικά μέτρα, δεν έχουμε μία ενιαία προσέγγιση παντού και όλα τα στοιχεία της πράσινης αρχιτεκτονικής είναι σημαντικά αν τα δούμε όλα μαζί, για να έχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας και θα εργαζόμαστε με έναν τρόπο πιο ολοκληρωμένο, με συνέργειες, με βάση τις υποχρεώσεις που έχουν τα κράτη-μέλη. Και έτσι η γεωργία θα χρησιμοποιείται περισσότερο για να ανταποκριθούν τα κράτη σε αυτές τις υποχρεώσεις, όπως είπα, για τα ζωτούχα, για τα ύδατα και για κάποια ε, φλαβερά στοιχεία τα οποία καταλήγουν στο χώμα. Σας ευχαριστώ. <coughs> Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Περνάμε τώρα στις παρεμβάσεις και ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Ράνς Γκαρσία, ε, για τους ηγητές δεν περιορίζουμε το χρόνο. Ιδιαίτερα, παρακαλώ. Κυρία Ράνς Γκαρσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σας ε, κύριε Επίτροπε και ευχαριστούμε θερμά για τις εξηγήσεις που μας δώσατε γιατί αυτό που μας είπατε είναι από τα πιο σημαντικά σημεία της πρότασης για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Είναι αλήθεια ότι το θέμα του, της οικολογικής αρχιτεκτονικής είναι πολύ σημαντικό. Το κεφάλαιο αυτό για, το, για την πράσινη αρχιτεκτονική έχει τραβήξει την προσοχή και της κοινή γνώμης αλλά και των γεωργών και κτηνοτρόφων εν ώψη της νέας μεταρρυθμίσης και είπατε κάτι που όντως ισχύει και θα πρέπει να εξασφαλίσει σε όλους μας ή να μας καθοδηγήσει, να μας κατευθύνει στο έργο μας. Θα πρέπει να εγγυηθούμε το μέλλον της γεωργίας. Όχι ε, γιατί είναι σημαντική η πλήρης απασχόληση, η καταπολέμηση της διάβρωσης του εδάφους, ε, η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά για όλο τον ευρωπαϊκό πληθυσμό έχει κρίσιμη σημασία να έχουμε γεωργία και κτηνοτροφία που σε προσιτές τιμές θα παρέχει ε, ποιοτικά προϊόντα και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το εξασφαλίσουμε για το μέλλον. Και στους περιβαλλοντικούς στόχους που κυρώσαμε στις διεθνείς συνθήκες ε, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και μια βιώσιμη γεωργία και κτηνοτροφία. Βιώσιμη και από οικονομική και από περιβαλλοντική άποψη. Θέλουμε φιλόδοξους, υπεύθυνους στόχους όπως είπατε, αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστικούς και όταν θα θεσπίσουμε τους δείκτες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θα πρέπει να είναι γνήσιοι και να λαμβάνουμε υπόψη ότι η γεωργία δεν είναι απομονωμένη στον κόσμο αλλά είναι μια επιπλέον οικονομική δραστηριότητα. Ε, μία από τις πολλές που έχει ο άνθρωπος και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Επίσης, η αιρεσιμότητα. Η προσπάθεια που κάνουν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τεράστια. Ήδη στην ισχύουσα ΚΑΠ. Ίσως κάπου κάναμε λάθος. Δεν καταφέραμε δηλαδή να πούμε στην κοινωνία πόσο τεράστια προσπάθεια, εργόδη προσπάθεια καταβάλουν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι. Γιατί η δική μα παραγωγή είναι η πιο υπεύθυνη στον κόσμο από περιβαλλοντική άποψη. Μόνο εμεί υποβάλλουμε στου γεωργού και κτηνοτρόφου μα τόσο υψηλέ περιβαλλοντικέ προδιαγραφέ. Και αυτό δεν το ε, προβάλαμε, δεν το εξηγήσαμε στου καταναλωτέ δεν το αναγνωρίσαμε δεόντως και δεν ξέρουν οι καταναλωτές που αγοράζουν ένα ευρωπαϊκό γεωργικό προϊόν τι τεράστια προσπάθεια αυτό ε, απέτησε από τους γεωργούς μας και τους κτηνοτρόφους μας. Χθες πολλοί Ισπανοί διάβασαν το πρωί μία μελέτη που έγινε ε, γιατί σε εισαγόμενα εσπεριδοειδή από τρίτη χώρα βρήκαμε 50 απαγορευμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ουσίες και παρόλα αυτά τα πορτοκάλια ε, κατάφεραν να διεισδύσουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Είμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι για αυτή την παράβαση. Θα πρέπει λοιπόν να εξηγήσουμε στην κοινωνία τι τεράστια προσπάθεια προϋποθέτει η ευρωπαϊκή γεωργία και εκτινοτροφία. Και δεν θα πρέπει να πνίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί η ενισχυμένη αιρεσιμότητα είναι ένα επιπλέον βήμα από αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε υποχρεώσει στους γεωργούς και κτηνοτρόφου που θα είναι όμως εφικτές και δεν θα τους οδηγούν σε μια οικονομική ασφυξία. Και επίση δεν θα τους ε, ε, δαιμονοποιούμε. Θα πρέπει να δώσουμε ενάψματα στους γεωργούς και κτηνοτρόφου να κάνουν ένα βήμα επιπλέον στις παραγωγές τους που θα πρέπει να εξακολουθούν να είναι ελκυστικές και προσοδοφόρες, να είναι και φιλοπεριβαλλοντικές και να καταλήγουν σε ποιοτικά προϊόντα για τον καταναλωτή και να αφήσουμε ένα περιθώριο ελιγμών. Και γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και το οικολογικό σύστημα για τον πρώτο πυλώνα και τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Θα πρέπει αυτά να είναι συμπληρωματικά, να μην επικαλύπτονται. Επίσης, ε, εγώ και οι σκιώδεις ηγητές ε, προσπαθούμε στα θέματα των στρατηγικών σχεδίων να καταλήξουμε σε συμφωνία που θα γίνει αποδεκτή από όλου και θα ευνοεί και τον κλάδο της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Και μια και θα περάσουμε και στη συζήτηση για τα οικονομικά, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να κατανείμουμε τα γεωργικά κονδύλια που δυστυχώς δεν θα αυξηθούν με δίκαιο τρόπο. Και φυσικά να μην συρρυκνώσουμε περαιτέρω το γεωργικό προϋπολογισμό και η κατανομή των κονδυλίων να γίνει από το πρίσμα του παραγωγού, του γεωργού και ένα σημαντικό τμήμα να τα αφήσουμε στις βασικές ενισχύσεις για τη βιωσιμότητα, γιατί αυτές συνδέονται με την εκπλήρωση κάποιων πολύ, περιβαλλοντικών, ε, πολύ απαιτητικών περιβαλλοντικών προδιαγραφών, που θα είναι ακόμη πιο απαιτητικές στο μέλλον. Και μάλιστα είναι προδιαγραφές που μόνο εμείς τις ε, πληρούμε στον κόσμο και αυτό θα φέρει σε πολύ δυσμενή θέση τους δικούς μας Γιώργους. Και ε, αν προσθέσουμε σε όλα αυτά και τις διεθνείς συμφωνίες, θα πρέπει να προσέξουμε και να μην θυσιάσουμε κλάδους ε, της ευρωπαϊκής παραγωγής. Επίσης, να λάβουμε υπόψη ιδιαίτερα ευαίσθητες παραγωγές. Για παράδειγμα, παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος, ε, εγωπρόβιος τομέας και προ... να είμαστε πολύ προσεκτικοί για τις περιβαλλοντικές μας απαιτήσει ε, Καλό είναι να λαμβάνουμε υπόψη τις αλλαγές από την διαφοροποίηση των καλλιεργειών στην αμυψησφορά. Ε, καλά, αλλά τι θα γίνει με την οριζοκαλλιέργεια που δεν έχει εναλλακτικέ ε, λύσεις. Να λάβουμε υπόψη λοιπόν αυτές τις ευαίσθητες παραγωγές που λόγω των διαπραγματεύσεών μας βρίσκονται σε δυσμενή θέση. Ε, για το ρύζι είδαμε ε, τι δυσκολίες δημιουργούνται για τους Ευρωπαίους παραγωγούς λόγω των μαζικών εισαγών από την Καμπότζη για παράδειγμα. Λοιπόν, θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την ευσυνείδητη προσπάθεια που καταβάλουμε όλες οι πολιτικές ομάδες και ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία μεταξύ μας. Πάντως, ε, καλό θα ήταν η πλειοψηφία της Επιτροπής Γεωργίας να δώσει το πράσινο φως σε ένα κείμενο και μια πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπής που θα είναι σε προσόφελος των Γεωργών, των ε, πολιτών αλλά και του περιβάλλοντος. Ο κύριος Αντρία, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη ε, για την καθυστέρησή μου έριξα μια γρήγορη ματιά στο έγγραφο και διαπίστωσα ε, τα βασικά του στοιχεία. Σας ευχαριστώ που ήρθατε καταρχήν κύριε Επίτροπε. Σίγουρα αυτή η πρόταση για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ε, είναι πολύ σημαντική. Και αυτή η πρόταση έχει τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι η ενισχυμένη ρεσιμότητα για τις άμεσες ενισχύσεις. Επίσης έχουμε περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα στο δεύτερο πυλώνα και ε, ένα τρίτο στοιχείο, ένα τρίτο άξονα που είναι το οικολογικό σύστημα που λαμβάνει υπόψη ε, τις ε, κλιματικές και περιβαλλοντικές απειλές. Οπότε έχουμε τρεις άξονες που μας οδηγούν φυσικά στο εύλογο ερώτημα του προϋπολογισμού. Έχουμε τα μέσα, τα απαραίτητα μέσα για να εξασφαλίσουμε αυτή τη μετάβαση που δεν είναι μόνο οικολογική και περιβαλλοντική, αλλά σφαιρική. Είναι πολλά τα διακυβευόμενα εδώ στη μετάβαση. Και ε, τα πρώτα δείγματα από το Συμβούλιο δεν είναι και πολύ εθαρρυντικά. Γιατί για το δημοσιονομικό σκέλος το Συμβούλιο είναι αδιάλακτο, αμετάκλητο. Οπότε πώς θα βρούμε ε, πόρους, γιατί ε, ακόμη και σταθερό προϋπολογισμό να έχουμε να μην μειωθεί και πάλι για να χρηματοδοτήσουμε τις νέες προκλήσεις ε, δεν έχουμε αρκετού πόρου. Οπότε, αν θέλουμε να ανταποκριθούμε και στι περιβαλλοντικέ προκλήσει και να το συνδυάσουμε με τι γεωργικέ προκλήσει, θα πρέπει από κοινού να προβλέψουμε τα απαραίτητα μέσα και πόρου. Και αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό εδώ. Βέβαια, απάντηση δεν έχουμε ακόμη. Αλλά είναι τόσε οι προκλήσει και, και οι νέε προκλήσει που λογικό είναι να προβληματιζόμαστε για τον προπολογισμό. Επίση, έχουμε και σε άλλες προκλήσεις που αφορούν πιο άμεσα τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αν η ευρωπαϊκή οικονομία πάει καλά, η γεωργική οικονομία πάει καλά, ε, σίγουρα η γεωργία είναι η πρώτη που προβληματίζονται για το περιβάλλον και το θέμα των τιμών βρίσκεται στο επίκεντρο του όλου προβληματισμού. Στην έκθεσή μου για την ΚΟΑ, την Κοινή Οργάνωση Αγοράς, προτείνουμε ένα νέο ρόλο ισχυρότερο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι ο τομεακό ρυθμιστή. Και όπω είπα και χθε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη μεγάλη αστάθεια των τιμών, τεράστιες διακοιμάσει στι τιμέ. Και αν είναι εξασφαλισμένο το γεωργικό εισόδημα, ο Γεωργό θα γίνει ενεργό παράγοντα και στην προσπάθεια για την περιβαλλοντική προστασία. Αλλιώ αν δεν έχουμε εγγύηση των τιμών θα έχουμε πρόβλημα. Επίση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το σκέλο λοιπόν τους μηχανισμούς διαχείρισης των κρίσεων και στις ρυθμίσεις για να δούμε τι θα γίνει με την αγορά, να υπάρξει ένα είδους ρύθμιση της αγοράς για να αποφύγουμε αυτή τη μεγάλη αστάθεια των τιμών. Επίσης, ίσως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε το ζήτημα της γενικότερης εμπορικής μας πολιτικής, γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Το θέμα του υπολογισμού, το θέμα των τιμών και το θέμα της εμπορικής πολιτικής ε, είναι συνειφασμένα και θα πρέπει να περιληφθούν σε ένα κοινό πακέτο, γιατί αν ο Γεωργός ε, θεωρήσει τα περιβαλλοντικά κριτήρια ως ε, περιορισμό του και υποχρέωση που τον ε, δεν είναι χειροπόδαρα, δεν μπορεί να συμμετέχει θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος, γιατί η γεωργία και το περιβάλλον ε, και το κλίμα φυσικά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη θέση του Γιώργου Και συμφωνώ με αυτά που είπε και η κυρία Γκαρσία προηγουμένως για τα στρατηγικά σχέδια. Ευχαριστώ κυρία Μίλλερ. Κύριε Επίτροπε, με συγχωρείτε που άργησα. Ήμουν σε μια γεωργική εκδήλωση χτες το βράδυ και συζητούσαμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Έχουμε πάλι εντατικές συζητήσεις ε, στη Γερμανία με τους αγρότες. Αλλά είμαι και σε επαφή με τα Υπουργεία και πραγματικά υπάρχει περισσότερη απελπισία παρά σαφήνεια αυτή τη στιγμή γιατί Μας λένε τα Υπουργεία ξεκάθαρα πως ε, θα πρέπει να υπάρξει τεράστια αύξηση των διοικητικών δομών ε, για να γίνει αυτή η αλλαγή με τις ετήσιες εκθέσεις ε, και αξιολογήσεις με στόχους δικτών, παραγωγής και αξιολόγησης. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί η τωρινή διοίκηση και σημαίνει αυτό θα έχουμε περισσότερη γραφειοκρατία. Για εμένα λοιπόν τίθεται το ερώτημα πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια απλοποίηση, πώς θα καταφέρουμε να έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια σε αυτόν τον τομέα. Ήδη έχουμε πολλές ε, τεχνικές συναντήσεις μεταξύ των σκιωδών εισηγητών. Μιλάμε για αποθεματικά κρίσεις, για γεωργικά αποθεματικά, αλλά στις λεπτομέρειες δεν προχωράμε. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και να μπορούμε να εξηγήσουμε στους αγρότες πώς ε, θα λειτουργεί αυτή η νέα γεωργική πολιτική και πώς ε, θα υπάρξει και κάποια απλοποίηση στην ε, διοίκηση. Στον λόγο σας μας εξηγήσατε το τι μας περιμένει. Θα ήθελα πραγματικά όλα όσα κάνουν κάθε μέρα οι αγρότες όσον αφορά το τοπίο, τα κοινωνικά ζητήματα, το περιβάλλον και το κλίμα να μπορούν να μπουν σε μια σχέση με την αιρεσιμότητα αυτήν. Αλλά αν ε, είναι τα πράγματα τόσο χονδροειδή όπως μας τα δείξατε τώρα, φοβάμαι ότι δεν υπάρχουν πια δυνατότητες στον δεύτερο πυλώνα για να έχουμε επιπρόσθετα εθελοντικά μέτρα. Και δεν ξέρω τι θα γίνει λοιπόν. Εγώ πάντα και οι φιλελεύθεροι ήμασταν ε, υπέρ ε, των εθελοντικών ε, μέτρων και να μπορούμε να παρουσιάσουμε έναν κατάλογο εθελοντικών μέτρων από τα οποία θα μπορούν να επιλέγουν οι αγρότες για να επιτύχουμε περισσότερα πράγματα για το κλίμα. Σας ε, παρακαλώ λοιπόν ε, πραγματικά να μας ε, ακούσετε και να συνεχίσετε να εξελίσσετε την πολιτική αυτή για τους καταναλωτές Ευρώπης, αλλά δεν χρειάζεται να περάσουμε σε απότομες τομές και μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας. Μάλιστα, ευχαριστώ. Όπως είπα στους εισηγητές μας δεν περιόρισα το χρόνο αγόρευσης. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους καλεσμένους κυρίες Αγγιλέρα από τον κλάδο των εσπεριδοειδών. Θα μιλήσουμε αργότερα για τα εσπεριδοειδή. Επίσης να καλωσορίσω και τους εκπροσώπους της ε, τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα περάσουμε τώρα στους συντονιστές. Οι συντονιστές θα έχουν περιορισμένο χρόνο αγόρευσης, δύο λεπτά. Πρώτα, ο κύριος Νταντάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Ευχαριστώ τον Επίτροπο που ήρθε. Πολύ εύστοχα μίλησε προηγουμένω η κυρία Ράζ Γκαρσία και θα ήθελα να το συμπληρώσω και από τη σκοπιά του ΕΛΚ. Είναι προφανέ ότι το θέμα του περιβάλλοντο είναι πολύ σημαντικό μα μέλημα και διακύβευμα και συμφωνούμε όλοι σε αυτό και οι Γεώργοι το ίδιο και οι κτηνοτρόφοι. Γιατί στην καθημερινή άσκηση τη γεωργική δραστηριότητα βλέπουν τι διαφορέ. Βέβαια, ε, νερό υπάρχει ακόμη, αλλά ανάλογα με την περιοχή τα έντομα δεν είναι τα ίδια όπως παλιά. Και υπάρχουν πολλές νέες συνθήκες που τους υποχρεώνει να κάνουν και αυτοί αλλαγές στη γεωργική και την κτηνοτροφία. Και οι στόχοι της κοινή γεωργικής πολιτικής, όπως φαίνονται στο άρθρο 39 της συνθήκης, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια των καταναλωτών, αλλά να εξασφαλίζει και το γεωργικό εισόδημα. Και δυστυχώ οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι στην περίοδο που πέρασε, καθ' όλη τη διάρκεια τη κοινοβουλευτικής μα θητεία και τη δική σας θητεία, δυστυχώς δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ικανοποιητικό εισόδημα σε όλους τους Ευρωπαίους αγρότε. Κάτι που δείχνει ότι οι δημόσιες πολιτικές μας δυστυχώς ε, πέτυχαν. Ήταν ε, ελλειπή. Και τώρα προσθέτουμε νέους περιορισμούς και νέες προϋποθέσεις. Αυτό ε, ε, θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους γεωργούς και κτηνοτρόφους, γιατί η γραφειοκρατία αυξάνεται και οι περιορισμοί το ίδιο. Και μάλιστα θα αποτρέψουμε νέους κυρίως γεωργούς να ασχοληθούν με τη γεωργική δραστηριότητα. Έχουμε δει στοιχεία για, τις, για την εξέλιξη της ε, κτηνοτροφής και της ειδικευμένης κτηνοτροφίας στην πατρίδα μου και για το 2018 είναι πολύ ανησυχητικά τα στοιχεία που λάβαμε γιατί φαίνεται ότι έχει καταρρεύσει η κτηνοτροφία, έχει μειωθεί το ζωικό κεφάλαιο, ε, έχουν καταποντιστεί πολλές κτηνοτροφικές μονάδες. Και αυτό είναι σημαντικό διακύβευμα της κοινής γεωργικής πολιτικής. Κυρία Νόιχλ, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Να με συγχωρείτε και εμένα για την ε, καθυστέρηση. Έχουμε και κάποια άλλα πράγματα που έπρεπε να κάνουμε. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Στηρίζω τις αρχές της πρότασης και θεωρώ ότι είναι σωστό να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε έναν θεμέλιο λίθο όπως είπατε ε, τον οποίο χρειαζόμαστε ε, ο οποίος θα συνδέεται ξεκάθαρα με τις οικολογικές ε, επιδόσεις. λυπούμε για το ότι δεν παραμείναμε στο εθελοντικό πλαίσιο Εγώ θα επιθυμούσα να ξεκαθαρίσουμε το ότι το δημόσιο χρήμα κυρίως θα πρέπει να δίνεται για παροχές ε, στην κοινωνία, δηλαδή για την προστασία του ύδατος, ε, της βιοπικιλότητας, ε, του περιβάλλοντος κτλ. Και ακριβώς αυτά στα οικολογικά αυτά σχέδια ε, παρατηρήσα ότι δημιουργούν τεράστια αβεβαιότητα στην ε, Γερμανία. Το σύστημα αυτό θα είναι επιτυχές ε, μόνο εάν μπορέσουν τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν κάποια προγράμματα για να τα εφαρμόσουν και πραγματικά εδώ πέρα ο συνάλφος από το ΕΛΚ, λυπούμε που το λέω, αλλά επιμένει ότι θα πρέπει 70% των πληρωμών του πρώτου πυλώνα θα πρέπει να πηγαίνει στο παραδοσιακό σύστημα άμεσων πληρωμών. Όχι, θα πρέπει να πηγαίνει ξεκάθαρα σε συνδεδεμένες πληρωμές ε, οι οποίες θα ωφελούν την κοινωνία και πρέπει να τα πείτε αυτά σαφώς. αυτό είναι νομίζω το βασικό πρόβλημα εδώ. Νίκολσον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν σκόπευα να πάρω το λόγο, αλλά σε κάποιο βαθμό ε, Όλοι αρχίσαμε να ανησυχούμε και μιλήσατε για 50% και όσοι δουλέψουν μέσα στην γεωργία τα επόμενα χρόνια θα πρέπει αυτό να το λάβουν υπόψη. Δεν υπάρχει αμφιβολία όπως είπε ο κύριος Νταντών ότι η γεωργία έχει αλλάξει. Τα ζώα είναι ακόμα έξω στη φάρμα μου, στη χώρα μου τώρα, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι μέσα είναι τόσο, τόσο, περισσότερο, τόσο πιο ζεστός ο καιρός. Υπάρχει, υπάρχουν πολλές αλλαγές, αλλά κάπως πρέπει οι γεωργοί να μπορέσουν να δουλέψουν ε, ε, τελικά, γιατί αυτοί είναι που εργάζονται 365 μέρες το χρόνο από το πρωί μέχρι το βράδυ και πρέπει και να αλλάξουν και να προσαρμοστούν στις νέες προκλήσεις. Επίσης είναι πολύ δαπανηρό όλο αυτό. γιατί υπάρχουν πολλά έξοδα. Και το τη γνώμη μου, πριν από καιρό έχω καταλήξει στο ότι οι Γεωργοί σε μεγάλο βαθμό έχουν αισθανθεί απόγνωση με τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται οι ευρωπαϊκοί κανόνες στα κράτη-μέλη. Και Ίσως αυτό θα πρέπει λίγο να το εξετάσουμε, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η ερμηνεία των κανόνων και η εφαρμογή είναι οι ίδιοι και δεν διαφέρουν από κράτος σε κράτος. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, πιστεύω. Ευχαριστώ. κυρία Κατάινεν. Äh, siitä, että uudessa CAP-esityksessä Σας ευχαριστώ. Εγώ πιστεύω πως η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ε, νέες συνθήκες να είμαστε κοντά στον κόσμο ώστε ε, ο κόσμος να νιώθει πως ε, καλύτερα λαμβάνονται αποφάσεις όταν είμαστε κοντά στον κόσμο. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό και φανταστείτε τον καιρό και τις διαφορές ανάμεσα στην Ισπανία και στη Φιλανδία. Οι διαφορές είναι τεράστιες. Ε, μείον 30 βαθμούς κάνει στη χώρα μου ε, αυτή τη στιγμή και κάπως έτσι θα είναι μέχρι τον Απρίλιο. Και βέβαια τα λοιπάσματα που χρησιμοποιούμε είναι διαφορετικά και πρέπει να ε, πληρούν διαφορετικές προδιαγραφές. Άρα λοιπόν, ποιες είναι οι δυνατότητες του κράτους μέλους να παρέμβει και να αποφασίσει για την κοινή γεωργική πολιτική. Ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι της Κομισιόν και πιστεύω πως τα κράτη-μέλη είναι σε καλύτερη θέση για να μπορούν να αποφασίζουν Πώς βλέπετε λοιπόν ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο, ο ρόλος, να αλλάξει ο ρόλος των ε, ε, κρατών μελών. Ευχαριστώ. Κυρία Σένερα. Ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, από τη δική μας πλευρά θέλουμε να επιμείνουμε ακόμα μια φορά πως είναι πολύ σημαντικό το να προσεγγίσουμε το πρότυπο παραγωγής, τη ρύθμιση των αγορών και τη ρύθμιση των τιμών. Ε, πολύ καλά είναι να συζητάμε για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, όμως το πρόβλημα είναι ότι διαρκώς μιλάμε για κάποια κομμάτια και για ε, μπαλώματα, αλλά η πραγματικότητα αλλού μας οδηγεί. Στην Γαλλικία έχουμε τεράστια κρίση λόγω της ε, μόλυνσης ε, που έχει προκληθεί λόγω των αποβλήτων από την βιομηχανική παραγωγή χείρων, ε, από τα χειροστάσια. Έχουμε λοιπόν ε, μια ολόκληρη γη η οποία έχει μετατραπεί σε χωματερή ε, και ρηπαίνονται και τα ύδατα. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε για πρότυπα, να μιλήσουμε για τιμές που εγγυώνται πως όλα τα άτομα τα οποία ασχολούνται με τη γεωργική δραστηριότητα και την κτηνοτροφία θα μπορούν να ζήσουν από την ε, δουλειά τους και αυτό συνδεδεμένο με ένα πρότυπο παραγωγής που πραγματικά θα αποφεύγει τέτοιες καταστάσεις περιβαλλοντικής κρίσης, ε, κρίσης τιμών και τελικά καταστροφής της υπαίθρου και των θέσεων απασχόλησης στη γεωργία. Σας ευχαριστώ. Κύριος Χόισλινγκ. Äh, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ας μιλήσουμε λίγο για την πραγματικότητα. Πώς θα λύσουν τα κράτη-μέλη τα προβλήματα τα οποία δεν λύσαμε εμείς στην τελευταία ΚΑΠ. Είναι λίγο αφελές. Η χώρα μου, η Γερμανία, έχει αυτή τη στιγμή 16 εκκρεμείς δίκες στο δικαστήριο για ζητήματα ΚΑΠ. Λοιπόν, αυτό το οποίο πρότεινε το Συμβούλιο είναι τελικά Δώσα μας τα λεφτά και κάτι θα κάνουμε και κατά προτίμηση εθελοντικά. Ε, έτσι δεν κάνουμε τίποτα και φαίνεται αυτή η αντίφαση και στις ε, προτάσεις σας. Ναι, εντάξει, λέτε χαμηλές τιμές, δηλαδή μαζική παραγωγή, ελεύθερο εμπόριο, εμπόδιο, εμπόριο με τις χώρες Μερκοσούρ, να κάνουμε εξαγωγές και μετά μας λέτε να φροντίσουμε και το περιβάλλον. Ε, δεν γίνονται αυτά. Χρειάζεται μια προστασία για να μην υφίστανται dumping οι αγρότες μας και από την άλλη όχι εθελοντικά μέτρα, αλλά υποχρεωτικά. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι δεδομένη ε, της δραματικής κατάστασης της εξαφάνισης των ειδών. Δεν μπορούμε να πειραματιζόμαστε κάνα δύο χρόνια να δούμε ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση, να δοκιμάσουμε αυτό και να δούμε τι θα γίνει. Η κρίση υπάρχει και πρέπει να λυθεί και είχαμε χτες και τους υπουργού. Ε, εντάξει το κλίμα είναι άφημα αλλά πείτε μας συγκεκριμένα μέτρα. Τι πρέπει να κάνει ο αγρότης για να έχουμε αυτή την εξοικονόμηση 40% στον τομέα του κλίματος. Δεν το βλέπω. Και είχαμε και διάφορες συνεδριάσεις ε, με την εισηγήτρια. Ναι, ε, δεν είναι δυνατόν συνεχώς να μειώνεται η απέτηση προς τα κάτω θα πρέπει και οι αγρότες να έχουν κάποιες προοπτικές ε, μακροπρόθεσμες ε, και τελικά να μην έχει την αίσθηση ο φορολογούμενος ότι τα λεφτά του πηγαίνουν κάπου γενικώ. χωρίς να υπάρχει καμία αλλαγή ε, του συστήματος που είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Σας... Ο κύριος Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το ελεγκτικό συνέδριο πρόσφατα συμπέρανε πω η περιβαλλοντική μα πολιτική δεν ήταν διόλου αποτελεσματική και μάλλον είπε τα είπε. Μάλιστα είναι τόσο ασυνεπής που, που βλάπτει, ζημιώνει τις ε, πιο προνομιούχες ε, εκμεταλλεύσεις ε, ενώ προσπαθεί να ευνοήσει μόνο που αυτές που κάνουν οικολογικές ή βιολογικές δραστηριότητες. Μια πρόσφατη μελέτη τοποθέτησε ωστόσο ότι η γαλλική γεωργία ανάμεσα στις πιο βιώσιμες του πλανήτη μπορεί να είναι ίσως αντίθετη με μάλλον Φαίνεται πως οι γεωργοί διαρκώς έχουν να αντιμετωπίσουν ε, καταστολή. Θα λάβετε υπόψη το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης των ευρωπαϊκών γεωργιών, προτείνοντας διαφοροποιημένες πολιτικές, ώστε να πάψει αυτή η, ο θέμητος ανταγωνισμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη και να ενεργήσουμε πραγματικά και αποτελεσματικά για το περιβάλλον. Και έπειτα, έχετε να πείτε για την εμπορική μας πολιτική, που στην ουσία καταστρέφει τις περιβαλλοντικές μας προσπάθειες, απλά μετεγκαταστεί τις, ε, τα προβλήματα. Ε, έπειτα ε, θα βάλετε στην Ευρωπαϊκή Γεωργία την πράσινη πολιτική ενώ θα μπορούσατε να προτείνετε ανταμοιβή όλων των περιβαλλοντικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι παραγωγοί. Νομίζω πως πολλά πρέπει να αλλάξουν. Αλλάξετε τη μορητική σας πολιτική που είναι πηγή μεγάλη σύγχυση υπέρ μιας πολιτικής κινήτρων που θα αναγνωρίσει επιτέλους τον υπεύθυνο ρόλο των γεωργών στη διατήρηση του περιβάλλοντος μας. Ευχαριστώ. Έχουμε 20 ομιλητέ που ζήτησαν το λόγο. Ένα λεπτό καθένας. Γιατί ο Επίτροπος δεν έχει απεριόριστο χρόνο, πρέπει σε λίγο να φύγει. Παρακαλώ να είστε πολύ συγκεκριμένοι και να θέτετε ερωτήσει, κύριε. Κύριε Αγγιλέρα. Καλώς. Επειδή με... έχω καλή ανατροφή θα πω μόνο καλημέρα, τίποτα παραπάνω. Σήμερα μιλούμε για τις ε, οικολογικές ενισχύσεις. Έχουν θετικά στοιχεία. Εγώ είμαι υπέρ του οικολογικού συστήματος, ε, το θετικό το μέτρο. Θα δούμε πώς θα το εφαρμόσουμε βέβαια. Αυτό που θα ήθελα να σας ε, διαβεβάσω και εκ μέρου των γεωργών, μάλιστα έχουμε μια ομάδα εδώ για τα σπεριδοειδή, ε, υπάρχει μεγάλη δυσπιστία και μεγάλη ανησυχία ε, μεταξύ των γεωργών και εκτινοτρόφων, γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει αμοιβαιότητα με, τα, με τις τρίτες χώρες για τα προϊόντα. Ούτε υπάρχουν κατάλληλα μέτρα αγοράς που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Ευρωπαίων γεωργών. Έτσι έχει η κατάσταση. Και αυτό που με προβληματίζει με τις οικολογικές ενισχύσει για να μην μακρηγορήσω, είναι και θέλω απάντηση. Πώς θα ελέγξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις πιθανές οικολογι... τους πιθανούς οικολογικούς φραγμούς, τους πράσινους φραγμούς στην εσωτερική αγορά, αν έχουμε διαφορετικό σύστημα για οικολογικές ενισχύσεις σε κάθε χώρα. Γιατί μπορούμε τέτοιου φραγμού οικολογικού να του έχουμε και εντό τη ενιαία αγορά, μια και θα είναι διαφορετικά τα αισθήματα που θα εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Πώ θα το αποφύγουμε. Σα ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε στις ε, δηλώσεις σας ξεκινήσατε με το ότι θέλετε να προωθήσετε την Ιφόρο ε, γεωργία. Συμφωνώ πραγματικά όσον αφορά τις προκλήσεις και αναμένετε, λέτε, υπεύθυνα σχέδια από τα κράτη-μέλη με βάση τις υφιστάμενες αναλύσεις. Το ερώτημα είναι ποιος θα κάνει τις αναλύσεις. Ε. Και αυτές, εξ όσων γνωρίζω, τα κράτη-μέλη τα κάνει. Ποιος τις ελέγχει τα στρατηγικά σχέδια αυτά αν το κάνει η Κομισιόν θα πρέπει να είναι πολύ λεπτομερής ε, αναλύσεις, αλλιώς δεν θα έχουμε καμία πρόοδο. Έχετε τις δυνατότητες λοιπόν στην Κομισιόν να κάνετε αναλύσεις ε, των 28 κρατών μελών και να τις ελέγξετε ώστε να δείτε πράγματι τα στρατηγικά σχέδια. Πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Δεύτερη ερώτηση για τα οικολογικά αυτά συστήματα. Ναι, μπορεί να αποτελέσουν ένα εργαλείο, αλλά πραγματικά τα αφήνεται εντελώς ε, στον εθελοντισμό και στην καλή διάθεση. Το ελάχιστο νομίζω, το είπε και στην Άλφος, είναι να πείτε πόσο τις 100 των πληρωμών θα πάει στις, ε, στα οικολογικά αυτά σχέδια. Αλλά οι αναλύσεις πρέπει να εξεταστούν σωστά για να έχουμε τα στρατηγικά σχέδια και να υπάρχει μια δέσμευση των χρημάτων με ένα συγκεκριμένο ποσοστό σας ευχαριστώ κύριο Σάγκη. Καλημέρα κύριε Επίτροπε, καλώς ε, ήρθατε και οπωσδήποτε καλωσορίζουμε την περισσότερη επικουρικότητα. Ε, μιλήσαμε για κλιματική αλλαγή και αν μιλήσουμε πραγματικούς επιστήμονες θα σας μιλήσουν για το ε, ηλιακό μήνυμο με ένας ηλιακός κύκλος που ξεκίνησε πριν από 150 χρόνια και πρέπει πράγματι να προσαρμοστούμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αυξήσουμε την γεωργία για να αντιμετωπίσουμε τον κρύο γερό, δηλαδή να αγκαλιάσουμε τα γεννητικά τροποποιημένα, ε, κάτι το οποίο δεν κάνετε. Μιλήσατε για την εξοικονόμηση των υδάτων, πράγματι πολύ αξιόλογο. Ε, υπάρχει πράγματι ένα σχετικό ε, φυτό το οποίο έχουμε στην Βρετανία ή μυδική, αλλά είναι ψυχανθές ε, ή από την άλλη πλευρά έχουμε το τριφύλι, το οποίο ε, εκλεί οξύδια του αζότου, πάλι και αυτό δεν σας αρέσει, τότε μπορεί να αυξηθούν οι αρωτρές ε, καλλιέργειες, γίνονται πιο αποτελεσματικές, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζονται νέες ε, τεχνικές. Τι θα κάνετε με αυτό, θα βάλετε μυρικαστικά, όχι γιατί αυτά εκπέμπουν μεθάνιο. Οπότε τι θα έχουμε μαζική ανεργία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ. Αν δούμε τα τελευταία χρόνια είναι σαν να μην ε, συνέβη τίποτα. Ο κύριος Χόισλινγκ άσκησε κριτική στο θέμα του ότι τα μέτρα αυτά είναι προαιρετικά. Αν δούμε όμως το ότι έχει γίνει στις ε, διαφορές περιοχές με τα αναπτυξιακά σχέδια. Π.χ. στη δική μου την περιοχή έχουν γίνει πολλά πράγματα στον τομέα της βιοποικιλότητας Έχουμε πάρα πολλά θετικά παραδείγματα αγροπεριβαλλοντικά. Αυτό το οποίο με ανησυχεί κάπως είναι ότι ήδη πέρσι είχαμε δει κάποια πράγματα τα οποία υπέστησαν μεγάλη κριτική όσον αφορά το λεγόμενο πρασίνισμα και τώρα έχουμε αυτό το πρόγραμμα δύο επιπέδων ε, και αποτελεί ένα επιπρόσθετο ε, πρόβλημα το οποίο δημιουργούμε. Δεν είναι ένα μοντέλο το οποίο θα πρέπει να καταργήσουμε το ιστάμενο μοντέλο. Είναι ήδη πολύ επιτυχημένο. Ο κύριος Κολομπιέ. Κύριε Επίτροπε, η διαπίστωσή σας και οι προτάσεις σας δεν είναι στο ύψος των προκλήσεων. Ο προϋπολογισμός του πρασινίσματος, μάλλον ο απολογισμός του πρασινίσματος είναι δραματικός. Καμιά έκθεση επίσημη και τίποτα το περισσότερο για τους γεωργούς. Οι μεγάλες ευθύνες φέρει η Κομισιόν. Τώρα υπόσχεστε να διορθώσετε αυτή την καταστροφή αφήνοντας περισσότερη ελευθερία στα κράτη-μέλη στην προσέγγιση τους στα περιβαλλοντικά μέτρα. Τα κατόφλια που ορίζεται στον πρώτο και δεύτερο πυλώνα ωστόσο είναι πολύ σημαντικά ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσει του περιβαλλοντικού και κλιματικού τη στόχους προβλέπει ότι 40% τη κοινή γεωργικής πολιτική θα συμβάλλει στο κλίμα και στο περιβάλλον. Πιστεύετε πραγματικά πώ οι γεωργοί μα θα δεχτούν να βλέπουν τόση βοήθεια να δίνεται στο περιβάλλον και στο κλίμα και σε ένα σωρό οργανισμούς και τόσο λίγα στι δικέ του συνθήκε ζωή που είναι όλο ένα και πιο δραματικέ, χωρί να υπολογίζουμε και την επιπλέον γραφειοκρατία για τα κράτη και για ποιο, με ποιο θα είναι το κόστος χωρίς να υπολογίζουμε και τους νέους κανόνες και νέο διοικητικό φόρτο στους όμους των γεωργών μας, ενώ εσείς μιλάτε για απλοποίηση. Ε, ε, τα κριτήρια για την χορήγηση αυτών των μέτρων από τα κράτη-μέλη δημιουργούν μια ακόμα πιο μεγάλη αβεβαιότητα νομική όσον αφορά την κατανομή των βοηθειών και των, των ενισχύσεων μάλλον και των όρων και προϋποθέσεων αντίθετα με τους γεωργούς ε, θα που, καλούνται να καταβάλουν ε, και τα ελάχιστότερα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως, ε, ενώ οι διάφοροι οργανισμοί δοτίζουν στη διάρκεια των ετών. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Συμφωνώ ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για το περιβάλλον. Έχω υποβάλει τις τροπολογίες μου για το 30%. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν φοβάμαι ότι τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Οπότε συμφωνώ για την επένδυση στο περιβάλλον. Αλλά κοιτάξτε, διαφωνώ με αυτά τα οποία ακούγονται στην αίθουσα. Οι νέοι αγρότες ε, τα παρατάνε με όλους αυτούς τους περίπλοκους ε, κανόνες. Ε, εισάγονται συνεχώς νέοι κανόνες, τους οποίους επινοούν οι διάφοροι περιβαλλοντικοί και δεν σκέφτονται καθόλου τους αγρότες όσον αφορά το προαιρετικό. Ναι, προαιρετικό, αλλά συνδεδεμένο με τα ε, λεφτά και σας παρακαλώ να υπάρχει και μια προβλεψιμότητα για τα επόμενα 7 χρόνια. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ροπέ. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, iš tikrųjų labai ačiū Jums, kad Jūs atėjote ir... Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Μας παρουσιάσατε αυτό το πρόγραμμα που είναι πολύ ενδιαφέρον για τους γεωργούς μας, οι οποίοι πολύ ανησυχούν για το τι ακριβώς θα μπορέσουν να κάνουν για να ευνοηθεί το κλίμα και το περιβάλλον. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν εξής. Οι απαιτήσει που βασίζονται στα νέα ε, σχέδια θα είναι τα ίδια για όλα τα κατημέλη. Ωστόσο, η στήριξη θα κυμαίνεται πολύ. Και ο αντίκτυπο του περιβάλλον είναι ο ίδιος παντού, σε κάθε χώρα. Άρα λοιπόν γιατί η στήριξη να εξακολουθεί να διαφέρει από κράτος σε κράτος. Εάν δεν καταφέρουμε τη σύγκληση δεν μπορούμε να μιλάμε για επιπλέον στήριξη ή για, συγγνώμη, για επιπλέον όρους. Ε, θα πρέπει να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Δύο ε, ερωτήσεις που μου κάνουν και οι αγρότες. Πρώτη ερώτηση για τους ε, δείκτες. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μετράνε και ο τρόπος ε, με τον οποίο θα γίνει αυτό διαφέρει από κράτος σε κράτος. Λοιπόν, η ερώτηση πώς θα μπορέσετε να συμβιβάσετε και να αποφύγετε τις διαφορές όσον αφορά τη μέθοδο μέτρηση και ποιος θα ελέγχει τους ελεγκτές. Δεύτερη ερώτηση, είπατε ότι θα έχουν περισσότερη ευελιξία τα κράτη-μέλη. Θα υπάρχει χώρος για μέτρα τα οποία δεν θα είναι συνδεδεμένα με την ε, παραγωγή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν κάποιος αλλάζει την ε, καλλιέργειά του και περνάει από την σόγια στην κράμβη, ε, ε, θα πρέπει να μπορεί να ανταμείβεται με κάποιον τρόπο. Τι θα κάνετε γι' αυτό, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, Επίτροπε. Και αυτή τη φορά μας διευκρινίσατε μία πολύ κρίσιμη περιβαλλοντική ε, ερώτηση και είναι κρίσιμη γιατί πρέπει να στηριχθούν όλοι οι Ευρωπαίοι ε, πολίτες ε, και άρα μεγαλύτερες φιλοδοξίες είναι βασικός στόχος. Όμως η δυσκολία είναι πώς θα βρούμε το μέσο όρο ανάμεσα στις περισσότερες φιλοδοξίες της γεωργικής πολιτικής ενώ ταυτόχρονα θα καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να επιβαρύνουμε περισσότερο με δυσκολίες τους γεωργούς λόγω περισσότερης γραφειοκρατίας. Φυσικά δεν θέλουμε οι γεωργοί να βγουν από την ΚΑΠ. Άρα λοιπόν ε, η ισορροπία ανάμεσα σε αυτά είναι πολύ ε, δύσκολη. Εσείς μιλήσατε για μια πρόταση για την μεταρρυθμίσή σας. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν είναι πώς θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε πως αυτή μας η δέσμευση, αυτή η δέσμευση μάλλον των κρατών μελών τελικά θα οδηγήσει σε μια λύση. Αυτή είναι η ερώτηση που σας υποβάλλω εγώ. Πώς μπορεί η Κομισιόν να βοηθήσει με κάποιο τρόπο, γιατί η περιπλοκότητα που μεταφέρεται στα κρατημέλη είναι μεγάλη. Σίγουρα. Πώς θα τα καταφέρουμε λοιπόν. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι εξαιρετικά λακωνικός. Κύριε Επίτροπε, και εγώ πιστεύω ότι τα μέτρα θα πρέπει να τα συντονίσουμε με τις ενισχύσεις που λαμβάνουν οι ε, γεωργοί στις χώρες μέλη. Γιατί δεν είναι σωστό ένας γεωργός που λαμβάνει 250 ευρώ στραματική ενίσχυση να τη χάνει ίση μεταχείριση με εκείνο που λαμβάνει 500 ευρώ ε, στραματική ενίσχυση. Θα πρέπει να προστατεύσουμε και τη γεωργία μας και τα το, τις γεωργικές εκτάσεις και θα πρέπει να εξασφαλίσω μια ισότιμη μεταχείριση. Έχουμε καταθέσει και τροπολογίες. Θα πρέπει να σκεφτούμε όλους αυτούς τους γεωργούς που είναι 42 και άνω χρονών και που δεν είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα στήριξη της γεωργίας, αλλά που παρόλα αυτά λαμβάνουν κάποια μέτρα για να προστατεύσουν τις γεωργικές εκτάσεις και την ύπεθρο και δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν στην αγορά οι άνθρωποι αυτοί αν δεν λάβουν ενισχύσεις είτε στα, στα πλαίσια του πρώτου είτε στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα. Κοιτάξτε τι γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείε. Εκεί έχουμε ένα νέο μοντέλο, το μοντέλο του νέου Γεώργου που επίσης λαμβάνει ενισχύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πώς γίνεται, Πώς ε, γίνεται να μην υπάρχουν ε, ε, στρεβλώσεις αγοράς και να έχουμε συγκρίσιμη κατάσταση σε όλες τις περιφέρειες και κοντά στα σύνορα, να μπορούμε να έχουμε συγκρίσιμες μετρήσεις επίσης. Επίσης κατάλαβα καλά ότι τα προϊόντα της δασοκομείας θα είναι επιλέξιμα για το μέλλον, γιατί ο ρόλος των δασών για την κλιματική αλλαγή είναι πολύ, πολύ σημαντικός για τη διατήρηση και τη γεωργικής πολιτικής. Έπειτα, στο δεύτερο πυλώνα θα διατηρήσετε αυτό που είναι ε, τα προγράμματα leader, που είναι τα πιο επιτυχή για την οικονομία μας και έπειτα πώς θα εξασφαλίσετε το ανάτοτα όρια, το κάπινγκ, πραγματικά ανάτοτα όρια με τις χώρες και τα Υπουργεία. Πολύ αμφιβάλλω αν θα τα καταφέρουμε και έπειτα καλωσορίζω τη δήλωση του ΕΛΚ ε, υπέρ της απαγόρευσης των εισαγωγών ε, από χώρες που δεν τηρούν κριτήρια όπως της Ένωσης. Ελπίζω πως αυτή η πλειοψηφία υπέρ της απαγόρευσης θα συνεχιστεί και αλλού και δεν θα μείνει μόνο σε αυτή την αίθουσα τώρα που έχουμε τους εκπροσώπους των εσπεριδοειδών. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Ντελαέ. Σας ευχαριστώ. Θέλω να επιμείνω ε, στο ότι αυτό που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει περισσότερο αν θέλουμε να αγγιηθούμε την αυτονομία μας στην ε, διατροφική είναι το θέμα της οικονομίας των γεωργών. Και δεν σας άκουσα να μιλάτε για διπλές επιδόσεις ε, τόσο οικονομικές όσο και περιβαλλοντικές στα μέτρα σας. Επίσης δεν άκουσα τίποτα για βιοοικονομία. Πιστεύω πως η γεωργία και η βιοοικονομία είναι στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να συσχετίσουμε. Μιλάτε για ένα σχέ... Μιλάμε για ένα σχέδιο για τις πρωτεΐνες, δεν άκουσα τίποτα να λέτε γι' αυτό ε, τη στιγμή που εισάγουμε σημαντικές πρωτεΐνες από άλλα μέρη του κόσμου ε, που οι Ευρωπαίοι δεν το θέλουν πια. Ε, αυτές, αυτά τα νέα χτυπήματα για τους γεωργούς δεν θα τα αισθανθούμε με τον ίδιο τρόπο η, παραγωγή άλλων περιοχών του κόσμου. Και έπειτα μιλήσατε για ε, απλοποίηση. Δεν πιστεύω πως αυτή η προσασή πρόταση είναι απλοποίηση για τους γεωργούς, ίσως για τη διοίκηση, αλλά όχι για τους γεωργούς. Ο κύριος ευχαριστώ πολύ. Για το ΓΕΑ 2 αναφέρατε την προστασία των γεών. Αυτό είναι θαυμάσιο και πρέπει να το κάνουμε, αλλά πρέπει να είναι και εφικτό. Η ε, ιδέα ότι θα πρέπει αυτό να είναι ένας βασικός όρος θα δημιουργήσει πρόβλημα. Εάν θέλετε να το επιτύχετε, πρέπει να αλλάξει από την κατάλληλη προστασία στη συντήρηση, η διατήρηση και έπειτα με ε, ε, ε, ενισχυμένους όρους να δώσουμε κίνητρα στον κόσμο για να προχωρήσουν σε αυτόν τον δρόμο. Αν θέλουμε να το επιτύχουμε πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την κατάσταση στην Ιρλανδία και η ιδέα ότι θα πρέπει αυτό να το κάνεις απλά και μόνο για τη βασική σου πληρωμή, όσο καλή ή κακή πιστεύεις ότι είναι, δεν πρόκειται να γίνει στην πράξη. Κάτι ακόμα, η αναφορά το μη παραγωγικό. Ε, εάν είμαστε σοβαροί για το ποια αγαθά θέλουν και μπορούν να προσπαράγουν παράγουν οι γεωργοί, πρέπει να διαγραφεί αυτή η ε, λέξη non-productive, μη παραγωγικό. Ε, για χρόνια η, τα έλη στην, στη χώρα μου ονομάζονταν μη παραγωγικά, όμως παράγουν τύρφη. Πώς μπορείς αυτά να τα λες μη παραγωγικά. Ευχαριστώ. Γενικώ. Ε, είμαι ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Γεωργία έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες ε, για να προφυλάξει το περιβάλλον. Βέβαια υπάρχει ένα σχίσμα μεταξύ πέθρου και αστικών κέντρων. Με το πρόγραμμα όμως για τα εξύπνα χωριά προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Η κατάσταση είναι δύσκολη για όσους μένουν στην Ήπεθρο και όσους ασκούν γεωργική δραστηριότητα. Υπάρχουν όμως σημαντικά προβλήματα ρήπανση του αέρα λόγω της εντατικής γεωργίας, ακόμη και στα χωριά, όχι μόνο στις πόλεις. Και στην Ανατολική Ευρώπη, δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι το νιώθουν αυτό το θέμα της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις ε, στο αυτό οικολογικό αρχιτεκτόνημα για να έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Καταρχήν θα πρέπει να προσχωρήσουν στον οικολογικό αυτό προσανατολισμό ή γεωργή. Δεύτερον, ε, θα πρέπει να έχουμε ε, μια κοινή στρατηγική, οπότε τα εθνικά στρατηγικά πλαίσια δεν ξέρω αν είναι συμβατά και επίσης να έχουμε απλούς ε, συμπληρωματικούς μηχανισμούς ε, και σαφείς. Και το θέμα της ενισχυμένης αρισιμότητας που είπατε, κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να προκαλεί υπερβολικές ρυθμιστικές υποχρεώσεις, γιατί ο σημερινός οικολογικός προσανατολισμός στηρίζεται στο σεβασμό των κανόνων και προκαλεί ελέγχους που είναι πολλές φορές ανέφικτοι για τις αρμόδιες διοικήσεις και που επιβαρύνουν τους γεωργούς. Θα πρέπει λοιπόν η αιρεσιμότητα να αποτελέσει ένα κοινό πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, για το πρόγραμμα αυτό των οικολογικών σχεδίων, θα πρέπει να φροντίσουμε ο μηχανισμός να είναι υποχρεωτικός για τα κρατη και ε, εθελοντικός για τους Γιώργους. Η κυρία Πετήρ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ τον Επίτροπο και να τον ευχαριστήσω για τις εξηγήσεις που μας έδωσε. Ε, το Κροατικό γεωργικό Επιμελητήριο είναι ένας οριζόντιος φορέας ε, στην Κροατία και θεωρεί ότι η νέα πράσινη αρχιτεκτονική θα πρέπει να αφορά μόνο τους ενεργούς γεωργούς και να αναγνωριστεί μέχρι τώρα συμβολή τους. Και η νέα πράσινη αρχιτεκτονική θα πρέπει να προβλέπει μεταβλητά επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς όμως να διακυβεύει ταυτόχρονα την ενιαία εφαρμογή. Επίσης, στόχος θα πρέπει, στόχος θα πρέπει να είναι η εξίσωση της ανταγωνιστικότητας που μπορεί να οφείλεται στο διαφορετικό βαθμό συμμόρφωση στα θέματα κλιματικών αλλαγών, προστασία του περιβάλλοντο και καλή μεταχείριση των ζώων. Επίση, θα πρέπει να έχουμε ισότιμη μεταχείριση των γεωργών σε όλη την Ευρώπη με τι νέε προτάσει, επιτρέποντα όμω ε, τι διαφορέ και τι ιδιαιτερότητέ του. Επίση, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο των μικροκαλλιεργητών, των μικρών γεωργών ε, και να ληφθεί υπόψη αυτό στο μοντέλο των ενισχύσεων για να μην τους επιβαρύνουμε υπερβολικά γραφειο, γραφειοκρατικά. Επίσης, ε, θα, δεν μπορούμε με την αύξηση των προκλήσεων να μειώνουμε ταυτόχρονα και τον υγειοργικό προπολογισμό. Θα είναι ανέφικτη εφαρμογή των μέτρων. Η κυρία Μαγκίνες, ευχαριστώ. Κύριε... Ευχαριστώ. Μπορείτε κύριε Επίτροπε να μου εξηγήσετε γιατί αποφασίσετε να τα αφήσετε προαιρετικά αυτά τα οικολογικά προγράμματα. Δεύτερον, κοιτώντας αυτό το διάγραμμα για την βιοπικιλότητα. Τι γίνεται όταν οι αγρότες έχουν αυτό το ελάχιστο 7% ή 10% γιατί αυτό το οποίο συνέβη στο παρελθόν είναι ότι οι αγρότες αυτοί αποκλείονται οπότε ενθαρρύνονται να ξεριζώνουν υφιστάμενους βιοτόπους για να τους ξαναφυτέψουν για να πάρουν την επιδότηση και ανησυχώ, δηλαδή συμβαίνει μαζικά. Μπορείτε λοιπόν να μας δώσετε μια εγγύηση ότι θα ζητήσετε από τα κράτη-μέλη να είναι πιο ευέλικτοι αντί για άκαμπτοι με αυτά τα μέτρα. Και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα της ε, μόλυνσης του νερού. Γνωρίζω πως ζητάνε οι γεωργοί συμβούλους για να κάνουν αυτά τα σχέδια. Θα υπάρξει λοιπόν ένας ολόκληρος κλάδος τώρα. Σας ανησυχεί αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ Μαρκ Θαραμπέλα. Τρεις Καταρχήν, ε, όπως είπε ο κύριος Νταντάν, θα πρέπει πρώτα να επαναφέρουμε ένα αξιοπρεπές γεωργικό εισόδημα για τους γεωργούς και τις αγρότησες ε, σε όλο τον κλάδο. Δυστυχώς υπάρχει έλλειψη γεωργικού εισοδήματος. Δεν υπάρχει ανταμοιβή δίκαιη για το έργο των γεωργών. Δεν θα πρέπει να κατηγορούμε εδώ τα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε και εμεί συνυπεύθυνοι, γιατί όταν ε, εγκρίνουμε νομοθετικά μέτρα, πάντα προσκρούμε στην πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε θα πρέπει να είμαστε συνεπεί στην ψηφοφορία με τι ιδέε μα. Και η απλούστευση επίση χρειάζεται. Πριν από 15 χρόνια, ήδη ο Στέφαν Λεφόλ μα μίλησε για την ανάγκη να περάσουμε από τον περιορισμό στι συμβάσει. Δεν θα πρέπει τα κράτη-μέλη όμω στη συνέχεια να περιπλέκουν τα πράγματα. Θα πρέπει να επαληθεύουμε την κατάσταση, να ελέγχουμε την ε, ε στάση των κρατών μέλων, να μην περιπλέκουν τα κράτη-μέλη και να κατηγορούμε μετά τι Βρυξέλλες. Επίση, θα πρέπει να συνδυάσουμε τη γεωργία με την περιβαλλοντική πολιτική, αλλά και με την αναπτυξιακή πολιτική και με τι εμπορικέ μα πολιτικέ διεθνώ. Να έχουμε συνάφεια μεταξύ των διαφορών πολιτικών, κάτι που δεν ισχύει σήμερα, ιδιαίτερα με την πολιτική για το ελεύθερο εμπόριο που εφαρμόζουμε. Ευχαριστώ. 10 και μισή πρέπει να τελειώσουμε κύριε Επίτροπε αυτή την ανταλλαγή απόψεων, οπότε ονονοητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τους βουλευτές. Να σας πω ότι το θέμα σήμερα αφορούσε το περιβάλλον, αλλά άκουσα και άλλες ερωτήσεις, θα τις απαντήσω όμως. Να απαντήσω αμέσως για τα χρήματα. Γνωρίζετε την οικονομική ε, κατάσταση και το τι συμβαίνει με το ΠΔΠ το Συμβούλιο αποφάσισε να αναβάλει την σχετική συμφωνία. προφανώς είναι μέρος αυτό της νομοθετικής διαδικασίας, αλλά βεβαίως ε, πιστεύω ότι, έχουμε, ότι αν έχουμε μια σοβαρή πολιτική για τη Γεωργία μπορούμε να ζητήσουμε και περισσότερα λεφτά για αυτήν. Και ένας τομέας που μπορεί να γίνει αυτό είναι να θεωρούνται μέρο της λύσης για το περιβάλλον και το κλίμα και την ποιότητα των υδάτων οι αγρότες. Και έτσι να έχουμε περισσότερους πόρους για τους αγρότες μας, για να έχουν μια πηγή εισοδήματος για οικολογικές υπηρεσίε και καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Κάποιοι λένε ότι θέμε πρώτα τα χρήματα πριν οριστικοποιήσουμε τα θέματα της ΚΑΠ. Είναι και αυτή μια άποψη, αλλά υπάρχει και η άλλη ότι όταν ζητάμε περισσότερα λεφτά πρέπει να μπορούμε να πούμε γιατί τα ζητάμε. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Λοιπόν, να σεβαστούμε σε αυτό. Νομίζω ότι όλοι στην ίδια πλευρά είμαστε. Θέλουμε να αυξήσουμε τους ε, πόρους ε, για τους αγρότες μας και συμφωνώ με τον κύριο Νταντών για αυτά τα οποία είπε για τα οικονομικά, αλλά η συνάντηση αυτή αφορούσε συγκεκριμένα το περιβάλλον. Βεβαίω και η οικονομική και η κοινωνική πτυχή είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Ε, και κυρία Ρέαν, βεβαίω όλοι συμφωνούν στο ότι η βιωσιμότητα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αν δεν είναι στην καρδιά τη πολιτική μα, δεν θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε του φυσικού πόρου για τι μελλοντικέ γενιέ. Και η αγορά επίση ε, το ζητάει αυτό. Να είναι η βιωσιμότητα στα προϊόντα τα οποία πουλάμε. Οπότε είναι συμπληρωματικά αυτά. Και ε, όλε οι συμφωνίε ελευθερου που συνάψαμε τελευταία περιέχουν ε, κάποιο επίπεδο προστασίας περιβάλλοντος ε, και για τις ε, τρίτες χώρες συγκρίσιμο με αυτό το οποίο έχουμε εδώ πέρα. Και δεν συμφωνώ με κάποια από αυτά τα οποία ακούστηκαν όσον αφορά το dumping τιμών. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, το ανέφερε ο κ. Χόσλινγκ. Εντάξει, ακούγεται ωραία, αλλά θέλουμε και στοιχεία για το αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ε, στείλτε μας και θα τα ερευνήσουμε αν υπάρχουν. Τέλος, ε, το έχω δει και για το ρύζι πρόσφατα, το οποίο περιληφθεί στην πολιτική τα πάντα εκτός ε, των όπλων. Για πρώτη φορά ακριβώς ε, για να βοηθήσουμε τους Ισπανούς και τους Ιταλούς αγρότες που ανησυχούν ιδιαίτερως για το dumping του προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Καμπότζη και τη Μαλαισία. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καλοδεχόμενο αυτό και δείχνει ακριβώς ότι ε, δεν έχουμε πρόβλημα να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στην διάθεσή μας ε, προς το συμφέρον των Ευρωπαίων αγορτών και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Και απέναντι σε διεθνή αντίσταση. Λοιπόν, κάνουμε πάρα πολλά για το περιβάλλον, ε, τα εργασιακά σε όλες τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου και στο Μερκοσύρου παραδείγματος χάρη δεν θα έχουμε συμφωνία εάν δεν τα επιτύχουμε αυτά. Επίσης αναφέραμε τον προπολογισμό και το περιβάλλον. Κοιτάξτε, δεν ανέβαλε η Κομισιόν τις ε, συζητήσεις, αλλά οι συζητήσεις για την κοινή οργάνωση αγοράς ε, βλέπετε εκεί πέρα πολλά καλά παραδείγματα όπου έχει λειτουργήσει ο κανονισμός αυτός. Η εμπειρία που είχαμε το 2015-2016 χρησιμοποιήσαμε πολλά μέτρα εκεί, τα οποία τελικά κατέληξαν σε μια σταθεροποίηση των τιμών για τους Γεώργους. Και στο ζήτημα επίσης της ε, αποθήκευσης ε, αποβιδωρωμένου γάλακτος ε, σε σκόνη και γιατί βεβαίω αλλάζουμε, όπως λέτε, μια συνταγή η οποία λειτουργεί τώρα, κυρία Ρουρ. Ε, δεν ξέρω με ποιον μιλούσατε εσείς στο Βερολίνο στην ε, Πράσινη Εβδομάδα. Εγώ μίλησα με τους Γερμανούς αγρότες και δεν ε, μου είπαν κάτι τέτοιο σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με αυτά τα οποία λέτε εσείς. Ξέρω πως κάποιοι σε κάποια κράτη-μέλη ανησυχούν ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο. Αλλά υπάρχει 50% μείωση του αριθμού των ε, δικτών και των αναφορών που θα κάνουν τα κράτη-μέλη σε σχέση με τώρα. Και ακριβώς εδώ πέρα ενσωματώνουμε τρεις πολιτικές σε μία. Υπάρχουν λιγότεροι δείκτες, αλλά είναι κοινοί Υπάρχουν ε, λιγότερες αναφορές, ε, υπάρχουν προγράμματα κινήτρων για τους γεωργούς μας. Είναι μια εθελοντική προσέγγιση. Οι έλεγχοι μειώνονται ώστε απαιτείται να έχει λιγότερο προσωπικό το γερμανικό κράτο. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει στα χωράφια. Υπάρχουν δορυφόροι πλέον, οπότε δεν ξέρω πού εκεί αυτό το οποίο λέτε ότι χρειάζεται περισσότερο προσωπικό. Ε, δεν νομίζω δηλαδή να ισχύει, αλλά αν ισχύει, δώστε μου κάποια εξήγηση. Ο κ. Νταντένα ανέφερε το ότι πρέπει να προσέξουμε το διοικητικό βάρος. Μόλις το απάντησα στην κυρία Μίλλερ, δεν θεωρώ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά για την ενίσχυση της ε, διατροφικής αλυσίδας. Νομίζω ότι εσείς ε, και άλλοι ακριβώς βοηθάτε τους ε, αγρότες στην θέση τους στην διατροφική αλυσίδα με το Omnibus κτλ. Λοιπόν, αυτές είναι κάποιες Αλλαγέ ε, τις οποίες προσπαθήσαμε να πετύχουμε πριν από χρόνια. Να υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία και οι κανόνε του ανταγωνισμού. Είχαμε την νομοθεσία για τις αθέμητε εμπορικές πρακτικές ε, και έχουμε και κάποιες προτάσει για την διαφάνεια της αγοράς. Οπότε θα είναι νομίζω ένα οικονομικό βήμα προς τα εμπρός, ε, όπως τονίσατε άλλωστε. Κύριε Μακλητά, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, το στρατηγικό σχέδιο της ε, ΚΑΠ δίνει κάποια ευελιξία στα κράτη-μέλη. Ξέρω ότι εσεί τα θέλετε όλα υποχρεωτικά, αλλά όσοι συναντάω, μη και όχι αγρότε, μου λένε ότι ε, η προαιρετική προσέγγιση είναι η καλύτερη. Αυτό μου λένε. Ε, στην διαβούλευση που είχα, αυτό μου είπαν όλοι. Και θεωρώ ότι αυτό ισχύει, αλλά πρέπει να φροντίσουμε τα κράτη-μέλη να δίνουν την ευκαιρία στου αγρότε μα να μπορούν ε, να κάνουν άλλες επιλογές όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος εάν αυτό επιθυμούν. Επίσης έχουμε τη μεταφορά του 15% από τον πυλώνα 2 στον πυλώνα 1 των κονδυλίων. Υπάρχει ευελιξία των κρατών μελών εάν αυτό επιθυμούν να υπάρχει περισσότερη περιβαλλοντική διάσταση. Υπάρχει ήδη αυτή η ευελιξία και την διατηρούμε. Η μεταφορά δηλαδή από τον ένα πυλώνα στον άλλον. Οπότε όσον αφορά την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου θα μπορούν να κάνουν περισσότερα τα κράτη-μέλη και να χρησιμοποιήσουν την ευελιξία μεταξύ των πυλώνων. Ξέρω το επιχείρημά σας για το 50%. Αυτό είναι ένα οικονομικό επιχείρημα, θα το συζητήσουμε μια άλλη μέρα, οπωσδήποτε θα μας απασχολήσει. Συμφωνώ με τον κύριο Νίκολσον ότι η ερμηνεία των κανόνων και η εφαρμογή των κανόνων έχουν τεράστια σημασία. Και η Κομισιόν πρέπει να λάβει εδώ πέρα τις ευθύνε τη για να μην έχουμε ακριβώ τα κράτη-μέλη να κάνουν υπερθεματισμό και να είμαστε και φιλόδοξοι για τον αγρότη. Θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα την προηγούμενη φορά και έχουμε διδαχτεί από αυτό. Και το ότι κάναμε ακριβώς 100 αλλαγές τα τελευταία δύο χρόνια στην απλοποίηση ε, δείχνει ότι ακριβώς οι απόψει σας ακούγονται όσον αφορά την εφαρμογή και την ερμηνεία αυτών των κανόνων. Θα συνεχιστεί αυτό και οι υπαλλήλοι εδώ πέρα θέλουν να βοηθήσουν. Κυρία Κατάινεν, πρέπει να γίνουν σεβαστε οι τοπικέ συνθήκε. Αυτό έχει ενσωματωθεί στην γενικότερη προσέγγιση και θα λάβει υπόψη τις πιο τοπικέ συνθήκε και ταυτόχρονα θα πρέπει να επιτευχθεί πάντα με σεβασμό στου εννέα στόχους. Έχουμε κοινού στόχου, κοινού δείκτες, κοινέ αναφορέ. Και εάν για κάποιο λόγο τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να εφαρμόσουν τα σχέδια τα οποία έχουν συμφωνήσει με την Κομισιόν, η Κομισιόν θα αναλάβει δράση. Και όπω κάνουμε αυτή τη στιγμή με τα σχέδια δράση και τι δημοσιονομικές διορθώσει, θα το κάνουμε ξανά για να επιτύχουμε τους ε, στόχους ε, τους πανευρωπαϊκούς, για να έχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού και ελάχιστες στρεβλώσεις το οποίο ανισχύει πολλούς ε, βουλευτές. Ε, κυρία Σένα, αν υπάρχει πρόβλημα με την ε, ρήπανση των υδάτων στην Γαλλικία από κάποια εκμετάλλευση με χείρινα, οπωσδήποτε δεν είναι υπόψη της Κομισιόν. Ενημερώστε το κράτος μέλος να εφαρμόσει την νομοθεσία. Δεν θα ασχοληθούμε με την μικροδιαχείριση σε επίπεδο περιφέρειας όταν υπάρχουν περιφερειακές αρχές, εθνικές αρχές και τα λοιπά Είναι ζήτημα επιβολής. Και αν μπορεί να βοηθήσει η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, ε, μια χαρά. Και Housing με κατηγορήσατε ότι είμαι αφελής. Ε, ίσως να είμαι. Ε, θα σας τα πει και ο κύριος Λάναγκαν Αλλά... Κοιτάξτε, τη τα συνδικάτα των αγροτών ε, και οι ΜΚΟ συναντήθηκαν, είχαν ε, μια πάρα πολύ καλή συζήτηση, αλλά δεν νομίζω ότι ό,τι και να πω εγώ για το περιβάλλον θα σας ικανοποιήσει, ό,τι και να κάνω. Οπότε εντάξει, ε, καταλαβαίνόμαστε. Αλλά εγώ θέλω να δώσω κάποια κίνητρα. Η δική σας προσέγγιση δεν λειτουργήσε αυτή η οποία είχε υποχρεωτικούς κανόνες και τα λοιπά και να δημιουργεί ένα κλίμα φόβου αγρότες για την εφαρμογή των κανόνων Αυτά είχαμε την προηγούμενη φορά και αναμένω τα στοιχεία για το dumping, το οποίο πάλι αναφέρατε, συχνά ακούγεται αυτό χωρίς καθόλου στοιχεία. Και Ελεσού, κάντε κάποιες ερωτήσεις ε, για την διαφορά στις πολιτικές. Εδώ πέρα επιμένουμε στους κοινούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχουμε κοινή πολιτική. Και θα πρέπει ακριβώς να μετράμε με κάποιον τρόπο το τι ε, συμβαίνει έτσι, επί τόπου. Για να ξοδεύουμε σωστά και τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Τώρα δεν θεωρώ ότι η εμπορική πολιτική καταστρέφει το περιβάλλον γιατί επιμένουμε όπως σας είπα σε διάφορες προδιαγραφές και θα συνεχίσει να ισχύει αυτό. Οπότε η περιβαλλοντική φιλοδοξία κατά την άποψή μου θα έλεγα μας βοηθάει για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Και έτσι πρέπει να το δούμε βεβαίως. Οι γεωργοί πρέπει να πληρώνονται για τα όσα κάνουν, για την παροχή δημοσίων αγαθών και για την διατροφική ασφάλεια, αλλά πρέπει να έχουμε και αξιόπιστες πολιτικές ε, στην πλευρά των δημοσίων αγαθών, ακριβώς για να ενισχύσουμε την θέση μας στις διαπραγματεύσεις του ΠΔΠ, για να έχουμε προπολογισμό για την κοινή γεωργική πολιτική. Οπότε είμαι υπέρ, όπως είπα, μιας ε, πολιτικής με κίνητρα. Κύριε Έγκλερ, συμφωνώ ότι η αμοιβαιότητα με τις τρίτες χώρες έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό το οποίο είπατε για τους ίσους όρους ανταγωνισμού σε σχέση με το περιβάλλον, όταν απομακρυνόμαστε από μια ενιαία προσέγγιση, πρέπει να έχουμε μια ισορροπία, όπως είπατε, για κάποια κοινά στοιχεία. Έχουμε κοινούς στόχους, λοιπόν, κοινούς δείκτες, κοινούς βασικούς κανόνες και δικλείδες ασφαλείας και κομψιών θα παρέμβει και θα παρεμβαίνει κάθε χρόνο για να εφαρμόζονται αυτά. Ε, υπάρχει μια ευελιξία στο σχεδιασμό των ε, προγραμμάτων. Και η κυρία Ντελα νομίζω ανέφερε την βιοοικονομία την οποία παραλείψαμε. Στην Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία νομίζω μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να έχουν εισόδημα οι αγρότες ε, και οι περιφέρειες. Και νομίζω είναι και καλή περιβαλλοντική πρακτική. Λοιπόν, είναι υποφελές για όλους. λοιπόν στην ανάλυση αυτή την οποία θα κάνει η Ισπανία για να δούμε τι θα γίνει για την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου για την ε, ΚΑΠ. Ε, εντάξει, γνωρίζω αυτά τα οποία λέτε. Έχουμε πολλές δικλείδες ασφαλεία όμως ε, για να υπάρχει μια κοινή εφαρμογή των πολιτικών. Κυρία Αλβερτή, η Κομισιόν θα διαχειριστεί ε, τους κοινούς στόχους, σας διαβεβαιώ. Έχω αναφέρει και την άποψή μου θεωρώ ότι η παρουσίαση που κάναμε για μια προσέγγιση με κίνητρα είναι η σωστή. Κύριε Άγνιο, με αναφέρατε τους ε, μόνιμους βοσκοτόπους, αλλά δεν ε, μου δώσατε συγχαρητήρια για το ότι καταργήσαμε τον κανόνα αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος είχε δυσαρεστήσει πάρα πολύ κόσμο και μας κόσε μάλλον κάποιους ψήφους, ε, γιατί τώρα υπάρχει και νομολογία πλέον για τις ε, χορτολιβαδικές ε, εκτάσεις αυτές και στον κανονισμό των Omnibus ε, έχουμε αντιμετωπίσει τις ανησυχίες μας και νομίζω φαντάζομαι θα συζητηθεί αυτό το θέμα τόσο ή άλλως. Και, Ντόφμαν, το ζήτημα το οποίο αναφέρατε και εσείς κύριε Πρόεδρε για την διπλή χρηματοδότηση και όλα αυτά τα ζητήματα το γνωρίζουμε. και ακριβώς προσπαθούμε να μην υπάρχει κάποια επανάληψη της ε, πολιτικής ε, και της ε, χρηματοδότησης. Κύριε Πρόεδρε, να μου ζητάτε να τελειώσω. Αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι τα θέματα τα οποία αφωνούν λεφτά, την μεταφορά μεταξύ διαφόρων πυλών θα συνεχιστούν. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποβάλουν σχέδια τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν. Τα κίνητρα αυτά, τα προγράμματα αυτά αποτελούν κίνητρο, θα έχουμε και την ε, δασοπονία η οποία θα περιληφθεί στο στρατηγικό σχέδιο, είναι στον πυλώνα 2 αυτή τη στιγμή, θα διατηρήσουμε το leader ένα 5% των χρημάτων και βεβαίως και η οροφή έχει μεγάλη σημασία, το πλαφόν, η προστασία, όπως ξέρετε, των υγροτόπων που απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα. Ξέρετε ότι εγώ το έκανα πάντα χωρίς την στήριξή σας, αλλά χαίρομαι που με στηρίζετε σήμερα. Ξέρω με ποιους συνεργάζονταν στο παρελθόν, τέλος πάντων. Οι ενεργοί αγρότες κτλ. και οι επαφές που ανέφερε ο κύριος Ταραμπέλα και οι εγγυήσει μας ε, για την βιοπικιλότητα είναι μέρος του στρατηγικού σχεδίου κυρία Μαγκίνες. Έχετε δίκιο λοιπόν, δεν θέλουμε να πάμε προς τα πίσω, κοιτάμε το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή και μετά θα είναι ένα στόχος που θα πρέπει ακριβώς να επιτύχουν τα κράτη-μέλη, να έχουν ένα σχέδιο για την βιοπικιλότητα. Οπότε ελπίζω οι ανησυχίες σας να μην ε, πραγματοποιηθούν τελικά και ακριβώ όπως σας είπα εμείς το κάναμε προαιρετικό γιατί σε αυτό πιστεύουμε είχαμε ένα υποχρεωτικό σύστημα, περισσότερου ελέγχου, περισσότερη ε, πολυπλοκότητα. Θέλουμε κάποια απλοποίηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους. Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να κάλυψα όλα τα ζητήματα. Θα ήθελα όμως ε, να σου πω ότι και ο κανονισμό τη ε, κοινή οργάνωση αγορά λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Σήμερα το πρωί συνεδρίασε η Επιτροπή όσον ε, αφορά την ε, σκόνη από βουτυρωμένου γάλακτος σε τιμή 1.158 ευρώ και άρα έχουμε πουλήσει 3 εκατομμύρια τόνους από σχεδόν 4 τα οποία ήταν σε αποθήκευση και βεβαίω όλα αυτά αντιμετωπίζουν την κρίση του κάλακτος και όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατά χωρίς την στήριξή σας. Ουσιαστικά έχει πολιθεί το 99% του αποθέματος, οπότε έχει λυθεί το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλό αυτό για το γάλα. Πολύ θετική είδηση. Ευχαριστούμε κύριε Επιτροπή για την ανταλλαγή αυτή απόψεων που ήταν απαραίτητη και για μας την Επιτροπή Γεωργίας. Αλλά πιστεύω ότι ήταν χρήσιμη και για σας αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Και φυσικά ήταν πολύ χρήσιμη και για τους συζητητές μας, γιατί έτσι θα επισπεύσουμε τις εργασίες για τις ε, διάφορες εκθέσεις. Γιατί δόθηκαν πολλές διευκρινήσεις, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστώ και θα σας δούμε και στο μέλλον. Προτείνω μια πολύ σύντομη, λιγόλεπτη διακοπή, τεχνική, να μπορέσουν και οι καλεσμένοι μας να πάνε για να να πιούν ένα καφέ γιατί θα έχουμε τουλάχιστον ένα μισή ώρα ψηφοφορία. Όποιο θέλει φυσικά δεν είστε υποχρεωμένοι, αλλά μπορείτε να πάτε να πιείτε ένα καφέ γιατί έχουμε να ψηφίσουμε σε λίγο. Δεν το Τέλος το διάλειμμα. Πρέπει να συνεχίσουμε. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον εισηγητή μας να λάβει το λόγο. Ε, Ο κύριος Ντόρμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συνέβαλαν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να μπορέσουμε να ψηφίσουμε σήμερα για να διαβιβάσουμε το ζήτημα στην, Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ λοιπόν όσους ε, διευκόλυναν την ε, επίσπευση των εργασιών ώστε να ψηφίσουμε σήμερα για να μπορέσουμε εμπρόθεσμα να περάσουμε στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Ψηφίζουμε 78 τροπολογία ε, διανοτάσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος, γιατί δεν σηκώσετε όλο καιρό στα χέρια. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 78, άρχεται ψηφοφορία. Μάλλον απορρίπτεται από ό,τι το βλέπω. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 80 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά απορρίπτεται 86 υπέρ κατά απορρίπτεται 84 υπέρ κατά απορρίπτεται 85 α, ηλεκτρονικός έλεγχος πρώτα για την 84 άρχεται η ψηφοφορία τέλος απορρίπτεται 85 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 2 της Επιτροπής Μεταφορών υπέρ, κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 1 της 5, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 ΠΕΤΗ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1. αρχιτή η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται, οπότε πάμε στην πρώτη τροπολογία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Εμβ υπέρ. Εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 106 υπέρ. Εγκρίνεται. 108 υπέρ. 108 υπέρ. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 108 άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 109 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 110 υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 109. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 110 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28 της ΕΜΒΗ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 118, 118 και σύναφης πανομοιότυπες. Μάλλον υπέρ κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για 118, 119 κλπ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. 120. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 121. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 136. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 22 της Επιτροπής Μεταφορών. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 139 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 140 υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 139 άρχεται ψηφοφορία. 139 έρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Αυτό είπαμε, 139, ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 140, ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 154. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 155. Υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 7, αρχιτεί ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 160, 160. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 160. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 160 έρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγώ είχα δει αρνητικό πρόσημο στο κατάλογο του ΕΛΚ στο κατάλογο ψηφοφορία. Εν πάση 166 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 8, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 22, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 167 υπέρ. 22, ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Κύριε Ντες, εγώ είχα θετικό πρόσημο στον κατάλογο ψηφοφορίας του ΕΛΚ. Πάμε στην 167 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εκτός μικροφώνου τα σχόλια. 167 Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εκατόν ενενήντα τέσσερα. 194. Ποιος είναι υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 175 και 176 πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες 175 και 176. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνονται 179 και 180. Ποιο είναι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. 181 υπέρ, κατά απορρίπτεται 182 και 183 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτονται 187 ποιος είναι υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται ψηφοφορία Τέλος. Απορρίπτεται. 184. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 185 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 186 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 188 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 189 υπέρ, κα, εγκρίνεται. 190 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 190, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος, απορρίπτεται. 192 και οι υπόλοιπε υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Συμβιβαστική 10, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 198 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Και πάμε στη 204. Και οι υπόλοιπες. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 204 και τις συναφείς. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνονται. Με μικρή διαφορά όμως. Τροπολογία 8 πέτη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20 πέτη. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 112. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 131. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 98. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογίε 7 και 4, ποιο είναι υπέρ, εγκρίνονται. 99 υπέρ, εγκρίνεται. 100 υπέρ, εγκρίνεται. 102 υπέρ, εγκρίνεται. 103 υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ, εγκρίνεται. Οπότε πάμε στη συμβαστική 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε στην 208, ε, ε, ε, συγγνώμη, υπέρ κατά εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 24 της ΕΜΒΗ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 212 υπέρ κατά απορρίπτεται 214 ή μάλλον πρώτο ηλεκτρονικός έλεγχος για την 212 άρχεται η ψηφοφορία τέλος εγκρίνεται 214 τώρα ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 215 υπέρ Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 214, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 215 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται, οπότε πάμε στην τροπολογία 226 και άλλες μαζί της. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία για τη 226 και τη συνάφης. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτονται ε, μία ψήφο διαφορά. Καλά που το ελέγξαμε. Τροπολογία 14 τραν υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 225 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 225. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 229. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 235 υπέρ κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. Zamykam głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μικρή διαφορά. 236. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 241 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 33 έμβη υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 34 έμβη υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 261, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 261, άρχεται η ψηφοφορία. Zamykam głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. 254. <laughs> Απορρίπτεται. 254 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 257 υπέρ. Κατά ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. μου. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. 248. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ζαμίκα. Τέλος. Απορρίπτεται. 251 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 244 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 244 άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 256 υπέρ. Εγκρίνεται. 252 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 200... Α, προηγουμένως να ελέγξουμε ηλεκτρονικά τις τροπολογίες 252 και 253 άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνονται. 247 και 249 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. εγκρίνεται. 246, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 250 υπέρ, εγκρίνεται. 245 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 315 υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται ψηφοφορία για την 315. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 262 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 258 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 263. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Με μία ψήφο διαφορά. 334 και οι υπόλοιπες μαζί υπέρ. Εγκρίνεται. 275 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 255 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε στην 266. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 21 της ΕΜΒΗ. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 278. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 243. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 288 υπέρ. Εγκρίνεται. 289 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 290 υπέρ. Εγκρίνεται. 291 υπέρ. Εγκρίνεται. 294 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 294. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 22 έμβη. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται 300 και λοιπές υπέρ κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 300 και τη συναφής. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. Τροπολογία 29. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 304. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 305 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 20 της έμβη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 20 της έμβη. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγγνώμη, λάθος. Ε, λέει ο πρόεδρος. Πάμε στην τροπολογία 6. Τραν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται. Τροπολογίες 259 και 260. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτονται. Συμβιβαστική 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 321. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 321. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με μικρή διαφορά όμω. 322 υπέρ. Εγκρίνεται. 323 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3... 32, συγγνώμη, υπέρ, εγκρίνεται. 325 υπέρ, εγκρίνεται. 326 υπέρ. Εγκρίνεται. 327 και λοιπές υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. 327 και συναφής. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μικρή διαφορά. 330 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικό έλεγχο για την 330 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. 329. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 331. Υπέρ? Εγκρίνεται. 332. Υπέρ? Εγκρίνεται. 333 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 333 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Παρατρίχα. 336 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 336 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 346. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 307. Υπέρ. Εγκρίνεται. 350 υπέρ. Εγκρίνεται. 240 και συναφής υπέρ. Εγκρίνονται. 12 της Επιτροπής Μεταφορών και άλλες υπέρ. Εγκρίνονται. Ηλεκτρονικός έλεγχος, γιατί το ζήτησε κάποιος ευρωβουλευτής, άρχεται η ψηφοφορία, τροπολογία 12 της Τραν και συναφής. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 312 υπέρ κατά απορρίπτεται. 314 υπέρ κατά απορρίπτεται. 104 και 10 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνονται. Τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 351 υπέρ. Εγκρίνεται. 352 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 353 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 της ΕΜΒΗ. Υπέρ. Εγκρίνεται. 311. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 355. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 356. Υπέρ. Υπέρ. 57 διορθώνει ο Κατά. Απορρίπτεται. 358 υπέρ κατά απορρίπτεται 359 υπέρ κατά απορρίπτεται 360 υπέρ κατά απορρίπτεται 361 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 361 άρχεται η ψηφοφορία τέλος εγκρίνεται. 362 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 362 άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 363 υπέρ. Εγκρίνεται. 364 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 365 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 20 άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στην 379 υπέρ κατά απορρίπτεται. 380 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 381 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 390. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 390. Τέλος εγκρίνεται. Συμβαστική 22. Ποιος είναι υπέρ, άρχεται η ψηφοφορία, συγγνώμη. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 391. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 392 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 400 υπέρ εγκρίνεται Συμβεβαστική 23 άρχεται η ψηφοφορία τέλος εγκρίνεται Συμβεβαστική 24 άρχεται η ψηφοφορία τέλος εγκρίνεται Πάμε στην 417. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία για την 417. Τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε στην 39. Ε, εγκρίνεται. Πάμε στην 31. Υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 25. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική 25. Τέλος. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 430. Άρχεται η ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 430 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 431. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ κατά απορρίπτεται 3 υπέρ ηλεκτρονικός έλεγχος για την 2 άρχεται ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 3 υπέρ εγκρίνεται τροπολογία 4 υπέρ Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την 5 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται με μικρή διαφορά. Συμβαστική 26. Άρχεται η, ψηφοφορία. άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τα 17 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Ε, εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά. διαφορά. 18. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Πάμε στην 25. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά. Απορρίπτεται. 27. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 28 υπέρ Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 28. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Για την 32. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 39. Ποιος είναι υπέρ κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 39 άρχεται ψηφοφορία. Τέλο Τέλος Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 42 υπέρ εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 43 άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 44. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 47. Ποιος είναι υπέρ? Ηλεκτρονικός έλεγχος πρώτα όμως για την 46 άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 46 λέει ο πρόεδρος. Λάθος. 47. 47 υπέρ κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 48 και 49. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 50 υπέρ. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται με το ίδιο αποτέλεσμα. 55, όχι 54 πρώτα. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά. 55 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία κατευθείαν ηλεκτρονικά. Τέλος. Απορρίπτεται. 56. Υπέρ. Εγκρίνεται. 57. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 30. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 64, δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 66. Πρώτο όμως ηλεκτρονικός έλεγχος για την 64, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά απορρίπτεται 71 υπέρ κατά απορρίπτεται 72 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία τέλος απορρίπτεται 74 υπέρ κατά Απορρίπτεται 75 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 76 άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 77 Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 77. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και ψηφίζουμε το σύνολο έκθεσης όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση όμως. Άρχεται η ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ο εισηγητής μας θέλει το λόγο μήπως, κύριε Ντόρμαν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ καταρχάς ε, για την έγκριση αυτής της έκθεσης σε επίπεδο της Επιτροπής. Δεν ήταν εύκολο, αλλά όλοι, ε, όλες οι πλευρέ προσπαθήσαμε να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις με του υπόλοιπου Και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συνεργάτες που δούλεψαν νυχθημερών για να ε, ολοκληρωθεί αυτή η έκθεση και για τα ζώα πρέπει κανείς να εργάζεται σκληρά και τώρα θα μπορούμε καλύτερα να τα υπερασπιστούμε. Οι μεταφορείς ε, οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι κτηνοτρόφοι το ίδιο. Δίνουμε ένα σαφέ μήνυμα στην Επιτροπή και στα κράτη-μέλη με αυτή την έκθεση με μια ώρα σειρά από συγκεκριμένα ζητήματα που απαιτούν πλέον δράση. Ε, Ευχαριστώ θα ήθελα, και μάλλον θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη στήριξη στη διάρκεια των εργασιών για, αυτή, για, για αυτό το φάκελο. Και όσον αφορά τις εξαγωγές προς τις τρίτες χώρες, περίπλοκο θέμα, πραγματικά μεγάλη μου χαρά που βρήκαμε συμβιβαστικές για όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ όλους και ευχαριστώ που μπορέσαμε να περάσουμε αυτή την έκθεση για την Ολομέλεια. Ευχαριστώ, ήταν πολύ σημαντικό που καταφέραμε και ψηφίσαμε την έκθεση αυτή, γιατί πάνω από 200 ευρωβουλευτές ζήτησαν τη σύσταση διερευνητικής επιτροπής και εμείς ζητήσαμε να παραμείνει στη δική μας αρμοδιότητα, τελικά τα καταφέραμε, έγινε, δεκτή, ε, έγινε δεκτό το αίτημα για καθήλια αρμοδιότητα της Επιτροπής μας, οπότε θα το διαβιβάσουμε πλέον στην Ολομέλεια το θέμα αυτό. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τους και οδησηγητές, τους βοηθούς, τους συνεργάτες τους, τη γραμματεία και να περάσουμε στο σημείο 10 για το οποίο έδωσε μάχη τόσο επιτυχημένα η κυρία Αγγιλέρα για να μπει στην ημερήσια διάταξη. Να έχουμε ανταλλαγή απόψεων με εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας για την κατάσταση των εσπεριδοειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθυστερήσαμε βέβαια κάπως τη συζήτηση λόγω της παρατεταμένης ψηφοφορίας. Ξέρουμε πώς έχει κατάσταση στην Ισπανία για τα εσπεριδοειδή. Ε, έχουν καταρρεύσει οι τιμές λόγω των πολύ ανταγωνιστικών ε, εισαγόμενων εσπεριδοειδών από τρίτες χώρες, από την Τουρκία, το Μαρόκο και μάλιστα στη μέση της ε, εσοδείας της περίοδου πώλησης. Θα μας μιλήσει ο κύριος Ζαόνο Φρέ εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της αγοράς περιδοειδών. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Σας ακούμε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Επιτροπή γνωρίζει τη δύσκολη κατάσταση της κατάστασης των εσπεριδοειδών στην Ισπανία στην πρώτο ήμιση αυτής της περίοδου. Θεωρούμε ότι συνδυασμό πολλών παραγόντων που κυρίω σχετίζονται με την παραγωγή στην Ένωση είχε αρνητικό αντίκτυπο στι τιμέ, ιδιαίτερα στην Ισπανία. Αυτό έχει να κάνει με την συγκομιδή τη ζήτηση, την ποιότητα του προϊόντος και τη διοργάνωση του τομέα. Την οργάνωση μάλλον του τομέα μεγάλη συγκομιδή. Ισπανική ε, καλλιέργεια φέτος θα οδηγήσει σε 13% μεγαλύτερη παραγωγή από την περασμένη περίοδο. Η δε παραγωγή των διαφόρων ποικιλιών συμπίπτει λόγω της ε, καθυστέρησης ε, ε, συγκεκριμένη συγκομιδή. Σε χαμηλή ζήτηση, ο κρύος καιρός συνήθω οδηγεί σε κατανάλωση φρούτων, όμως ε, το φθινόπωρο ήταν ιδιαίτερα θερμό και γι' αυτό δεν υπήρξε μεγάλη ζήτηση, άρα μείωση των τιμών. Ποιότητα. Η παρατηρημένη καλοκαιρινή περίοδο και η εκθυρασία οδήγησε σε μικρό μέγεθο των καρπών στι αρχέ τη περίοδου και άρα χαμηλότερε τιμέ. Επιπλέον, οι μεγάλε βροχοπτώσει και πλημμύρε τον Οκτώβριο επιδίνωσαν ακόμα την κατάσταση και αποδυνάμωσαν και άλλο τη ζήτηση. Έπειτα, πολύ χαμηλό επίπεδο οργάνωση αγορά. Ο τομέα των δεν χαίρει μεγάλη οργάνωση. Αυτό που είναι σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση, κατά τη γνώμη μα, είναι να τονίσουμε λόγοι δεν, σε ποιου λόγους δεν οφείλεται η κρίση. Η Κομισιόν δεν έχει καμία απόδειξη ότι η δύσκολη κατάσταση της αγοράς οφείλεται αποκλειστικά στην εισαγωγή από τρίτες χώρες, ιδιαίτερα από την Νότια Αφρική και την Αίγυπτο. Οι εισαγωγέ από την Νότια Αφρική ήταν 5% ψηλότερε από ό,τι το 2017. Ωστόσο, οι εισαγωγέ στη διάρκεια της περίοδου που καλύπτεται από την εκχώρηση ήταν πολύ χαμηλότερες. Ε, επίσης δεν υπάρχουν ενδείξεις από ότι η Βόρειος Αφρική μπορεί να είχε ε, επιπτώσεις στην Ισπανική περίοδο γιατί οι εισαγωγές ξεκίνησαν μόνο το Δεκέμβριο και φτάνουν στην αιχμή τους τον Απρίλιο. Οπότε η κατάσταση της αγοράς προκύπτει από συγκεκριμένες εσωτερικές ε, συνθήκες της παραγωγής. Άρα η εφαρμογή των ασφαλιστικών μέτρων σε σχέση με τις αγωγές δεν αιτιολογείται. Η Κομισιόν φυσικά θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα προϊόντα τα εσπεριδοειδή ε, για να διαπιστώσει οποιαδήποτε πιθανή διαταραχή για την, αγορά, για την ευρωπαϊκή αγορά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχουμε τον κατάλληλο χρόνο για τη συζήτησή μας. Εγώ θέλω καταρχάς να πω ότι δεν πρόκειται για ισπανικό πρόβλημα. Τα εσπεριδοειδή της Βαλένσιας και της Ανδαλουσίας και οποιοδήποτε πρόβλημα ε, των εσπεριδοειδών είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Είναι αλήθεια ότι έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή στην Ισπανία, αλλά δεν είναι πρόβλημα της Ισπανίας να πω αυτό στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, γιατί εάν το περιορίσουμε στην Ισπανία δεν προχωράμε καλά. Έχουμε λοιπόν διάφορες περιστάσεις, φυσικά υπάρχουν προβλήματα, δεν το αρνούμε εφόσον είναι προφανή, υπάρχει πρόβλημα της ε, ε, συγκομιδής, είχαμε αντίξωες κλιματικές συνθήκες, είχαμε περίοδο ξηρασίας και μετά πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις ε, που ε, οδήγησαν σε προβλήματα στα μεγέθη των εσπεριδοειδών Και τα προβλήματα αυτά συνέπεσαν, όμως θα πρέπει να σας πω να, να υποβάλω μόνο μια ερώτηση στον πρόσωπο της Κομισιόν. Πέρα από το εξηρασία, ε, κάθε φορά ε, συμπίπτει ο χρόνος της ε, περίοδου ανάμεσα στο νότιο και στο βόρειο ημισέριο και αυτό οδηγεί σε προβλήματα και μάλιστα με τη νέα συμφωνία που είχε μεγάλη ε, επιρροή φέτος είναι ότι αυτές οι έξι εβδομάδες παράτασης των πιο μικρών ε, αγροκτημάτων από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου δεν βοήθησαν αντίθετα επιδείνωσαν την κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια ε, αυξάνονται οι εισαγωγές από τρίτες χώρες. Ναι, βεβαίως δεν είναι μόνο η Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική, η Αίγυπτος, η Τουρκία. Με την Νότια Αφρική η κατάσταση είναι ιδιαίτερη γιατί ε, δεν θελήσατε να το σκεφτούμε. Υπάρχει μία ενδυμική πληγή. Είναι το μαύρο στίγμα που επιτρέπει να εισάγονται προϊόντα όπου έχουν μειωθεί οι απαιτήσει. Και οι εισαγωγέ αυτών των προϊόντων σημαίνει πως έχουμε μεγαλύτερη ε, παραγωγή η Νότια Αφρική. Αυτά τα θέματα, όπως σας είπα, δεν είναι μόνο η Νότια Αφρική, είναι και άλλες χώρες όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία. Έχουμε λοιπόν σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια εισαγωγών. Πώς είναι δυνατόν να αυξάνονται οι εισαγωγές από τρίτες χώρες, όχι μόνο την Νότια Αφρική, 5% είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ποια είναι η αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες γενικώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε τι κερδίζουν οι γεωργοί της Βαλένσια, της Αδαλουσίας, οι Ευρωπαίοι γεωργοί. Δέκα, δέκα ε, λεπτά όλα και όλα. Πέρυσι είχαμε τον ίδιο μέσο όρο για τα πορτοκάλια όπως και πριν τρεις δεκαετίες. Έχει μείνει σταθερό. Δηλαδή αυτό πια ε, δεν γίνεται. Το είπα και το αναγνωρίζω ότι υπάρχουν προβλήματα στον τομέα, ότι πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα, όμω το κλίμα δεν περνάει από τα χέρια μα. Να βελτιώσουμε τη δομή, ναι, βεβαίω, στην ΚΟΑ, αλλά υπάρχουν άμεσε επιπτώσει των εισαγωγών στην Ευρώπη με τη μείωση της παραγωγής των εσπεριδοειδών και, των χαμηλ... και τις χαμηλές τιμές. 10 λεπτά ε, το πορτοκάλι. Το κιλό, το πορτοκάλια. Ε, ε, δεν είναι λογικό τέτοιο, κάτι τέτοιο και ούτε είναι πρακτικό. Έχουμε λοιπόν αύξηση των εισαγωγών από την Νότια Αφρική και από άλλες χώρες. Πρέπει λοιπόν να δούμε το 2026 ε, θα απελευθερωθούν οι αγορές των σπεριδιδών και ο Επιτρόπος σήμερα το προείπε ότι πρέπει να υπάρχουν πολύ ψηλές απαιτήσει όσον αφορά την υγειονομική προστασία και την παραγωγή. Αυτό δεν συμβαίνει με τις τρίτε χώρε. Δεν υπάρχει αμοιβαιότητα όπως θα έπρεπε. Άρα λοιπόν, έχουμε κόστος παραγωγής πολύ ψηλό, όπως απαιτεί η ευρωπαϊκή κοινωνία, αλλά δεν το απαιτούμε από τις τρίτες χώρες τις ίδιες ε, προϋποθέσεις. Δεν παράγουμε τις ίδιες οι Ευρωπαίοι και οι Νότιο Αφρικανοί. Είναι διαφορετικές οι απαιτήσει και άρα δεν υπάρχει αμοιβαιότητα. Και εφόσον δεν υπάρχει αμοιβαιότητα, υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Υπάρχει dumping. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να, θέλω, να, μην, να κάνουμε όπως δεν βλέπουμε και να αφήνουμε να φτάσει το 2026 και να τελειώσει ε, τα, να τελειώσουν τα πορτοκάλια και οι Ισπανοί και οι Ευρωπαίοι Γεωργοί. Δείτε ποιε είναι οι επιπτώσει αυτών των εισαγωγών, γιατί αυτό που θα εξαφανιστεί είναι οι γεωργίε περιοδοειδών στη χώρα μου. Και εμεί αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Σα ευχαριστώ, κυρία Σένερ έχει το λόγο. Και εσείς απεριόριστα μπορείτε να μιλήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι κατά τη γνώμη μου είναι κοινικό, για να μην πω προσβολή στη νοημοσύνη μας, να έρχεστε και να μας λέτε ότι το πρόβλημα των χαμηλών τιμών σπεριδοειδής στην Ισπανία οφείλεται σε τεχνικά ζητήματα και σε θέματα παραγωγής ή έλλειψη οργάνωσης των παραγωγών. Ε, είδατε πού καταντήσαμε. Εγώ θα έλεγα ότι το πρόβλημα είναι πολιτικό. Ένα πολιτικό πρόβλημα που συνεχίζεται εδώ και χρόνια και πέφτουμε συνεχώς στην ίδια παγίδα. Ε, για όλα αυτά είναι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που τόσο ε, χαρούμε να συζητούμε και εγκρίνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς τη δική μου ψήφο φυσικά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γυρίσουμε λίγο πίσω, να πάρουμε απόσταση και να αναγνωρίσουμε ότι η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών είναι μια παταγώδης αποτυχία. Θα πρέπει να το παραδεχτούμε, γιατί το μόνο που θα πετύχουν είναι η καταστροφή της μικρομεσαίας γεωργίας και των μικρομεσαίων καλλιεργητών στην Ευρώπη και στις χώρες που συνυπογράφουν τις συμφωνίες μαζί μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να θελοτυφλούμε έχουμε την ευκαιρία να διορθώσουμε την κατάσταση με τη νέα κοινή γεωργική πολιτική, που όμως εξακολουθεί με τη μορφή που έχει τώρα να δίνει έμφαση στη γεωργία της εξαγωγής και έμφαση στις διεθνείς ε, συμφωνίες και, εμπορικές, και το ελεύθερο εμπόριο. Σήμερα ε, είναι η παραγωγή, αύριο θα είναι η γαλακτοπαραγωγή, την επαύριο η παραγωγή ε, βοήου κρέατος. Πότε θα σταματήσει αυτή η κατάσταση με τις κρίσεις, πότε θα σταματήσει ε, αυτή η εμπιστευτικότητα γύρω από τις διαπραγματεύσεις, τι συνέπειες θα έχουν οι εμπορικές συμφωνίες που συνάπτεται ε, για τους Ευρωπαίους γεωργούς. Θα πρέπει όλα αυτά να τα σκεφτούμε πολύ σοβαρά, παρακαλώ. Ο κύριος Κολομπιέ. Κύριε Πρόεδρε, Ακόμα μια φορά η κακή διαχείριση των ε, των ε, δικών μας παραγωγών απέναντι στις εισαγωγές από τρίτες χώρες είναι, δείχνει ακόμα μια φορά καταστροφική. Είναι σκανδαλώδης η η μεταχείριση αυτών των ε, ανθρώπων. Αυτή τη φορά είναι οι Ισπανοί και τα σπεριδοειδή. Φυσικά και η Γεωργία θα έπρεπε να είναι και όσια λόγω της ευαισθησίας της και του αντικτύπου της στην, ε, ε, στο περιβάλλον να μην υπάρχουν εισαγωγές σπεριδοειδών στη διάρκεια της εποχής τους και το ίδιο και για τα υπόλοιπα προϊόντα. Να μην υπάρξουν Ε, να μην γίνουν κρυζώσει, κάτι τέτοιο θα ήταν παραπετρελό. Ε, στην Φλόριδα υπάρχει ε, επίσης αυτό το φαινόμενο για να καταπολεμηθεί αυτό το, τα μαύρα στίγματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση απειλούνται εκατοντάδες ε, δέντρα ε, ελήψη κατάλληλης εμπορικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρτσελεζή. Μαρτσελεζή. Eh, Ευχαριστώ. Και με θλίβει αλλά και με εκνευρίζει ιδιαίτερα η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στη μεγάλη δυσαρέσκεια που υπάρχει ε, στους Ισπανούς κυρίους Γεωργούς με θλίβει και με εξοργίζει ταυτόχρονα η απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί χωρίς καμία απολύτω αυτοκριτική, χωρίς καμία συνέστηση, καμία συμπαράσταση και συμπόνια προ τους Γεωργούς, ε, δεν ξεκινά καν να σκέφτεται να λύσει το πρόβλημα. Αγανάκτηση υπάρχει και στην Ισπανία, στη Βαλένσια, πάνω σε πάνω από 50 οργανώσεις έχουμε διαμαρτυρία και μας ακρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καταποντίζονται οι τιμές. 14 λεπτά το κιλό το πορτοκάλια πληρώνουν, ενώ το κόστος παραγωγής είναι 20 λεπτά το κιλό διατίθενται σε τιμές κάτω του κόστους. Αυτή είναι η κατάσταση στα χωράφια της Ισπανίας, στα χωράφια της Βαλένθια, στους οπορώνες ε, της Ισπανίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, δεν μπορούμε να φλούμε. Έχουμε τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Νότια, με την Αφρική. Και δυστυχώς με αυτή τη ε, συμφωνία με την ε, Νότια Αφρική η η Νότια Αφρική μπορεί να εξάγει αδασμολόγητα εσπεριδοειδή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι το 2026 θα πληρώσει ούτε ένα ευρώ δασμό. Και μάλιστα αυτά τα όψιμα πορτοκάλια ε, και τα πρόωρα δικά μας θα συμπέσουν στις αγορές με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν οι τιμές. Και θα σας δώσω ένα στοιχείο για να καταλάβουμε, γιατί καλά τα ποσοστά, αλλά αν τον Οκτώβριο του 2016 η Νότιος Αφρική εξέγεγε 54.000 τόνους ε, πορτοκάλια, τον ίδιο μήνα του 2008 ήταν 142.000 οι τόνοι εξαγωγών. Τριπλασιάστηκαν οι εξαγωγές της ε, πορτοκαλιών της Νοτιού Αφρικής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενώ, ενώ εμείς και δικαίω, γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε την υγεία των καταναλωτών μα. υποχρεώνουμε όμω του δικού μα παραγωγού να τηρούν αυστηρότατε φυτογεωνομικές, κοινωνικέ και περιβαλλοντικέ προδιαγραφέ, τι γίνεται στην Νότια Αφρική. Έχουμε έναν απόλυτα αθέμητο ανταγωνισμό. Τελείω αθέμητο ανταγωνισμό ανταγωνισμός των προϊόντων της Αφρική. Και μάλιστα έχουμε μια σημαντική μια κυβερνητική οργάνωση της Βαλένθια που μας υπενθυμίζει ότι οι παραγωγοί της Νοτιοαφρικής χρησιμοποιούν στα, στα εσπεριδοειδή τους πάνω από 50, και το τονίζω, πάνω από 50 απαγορευμένες δραστικές ουσίες φυτογειονομικών προϊόντων. Εμείς έχουμε απαγορεύσει, ενώ εισάγουμε προϊόντα από τρίτες χώρες που τις χρησιμοποιούν. Υποτίθεται ότι συνάπτουμε συνθήκες για να βοηθήσουμε τις χώρες του Νότου και έχουμε ένα, μια μελέτη για την, για Νότια Αφρική που μας βεβαιώνει ότι μόνο το 2% των εξαγωγέων ε, πορτοκαλιών από την Νότια Αφρική είναι μαύροι. Οι υπόλοιποι είναι λευκοί μεγαλογεοκτήμονες. Οπότε δεν στηρίζουμε με τις εμπορικές συμφωνίες ούτε τους ντόπιου παραγωγούς, ούτε τους μικροπαραγωγούς που χρειάζονται τη βοήθειά μας στην Νότια Αφρική. Οπότε ανακύπτουν πολλές ερωτήσεις και με αυτές θα τελειώσω με ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Γεωργίας. Πρώτον, γιατί η Επιτροπή Γεωργίας δεν ενημερώθηκε για τι διαπραγματεύσει ε, για την εμπορική συμφωνία με την Νότια Αφρική, γιατί δεν δόθηκε γνωμοδότηση από την Επιτροπή μα όπω θα έπρεπε για τη συμφωνία αυτή και αν η ΚΑΠ θεωρεί ότι ένα από του στόχου τη είναι να εξασφαλίσει αξιοπρεπέ γεωργικό εισόδημα για του γεωργιούς, γιατί επιτρέπουμε ε, εισαγωγή προϊόντων που δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό και καταποντίζουν τις τιμές Επίση, Επίσης αναφέρεται ότι η ΚΑΠ θα πρέπει να εξασφαλίζει για τους Ευρωπαίους ε, ασφαλή τρόφιμα και ποιοτικά. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν με τέτοιους στόχους να επιτρέπουμε να εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα στα οποία έχουν εφαρμοστεί δραστικές ουσίες και φυτοφάρμακα που εμείς έχουμε απαγορεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά. Ευχαριστώ και πιστεύω ότι θα πρέπει να εγγύψουμε στο βαθύτατο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτό το μη βιώσιμο και ιδιαίτερα άδικο σύστημα που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί η Νότιος Αφρική και οι εισαγωγές της είναι μόνο η, κορυφή του παγόβουνου. Έχουμε πορτοκάλια από την Αίγυπτο, το Μαρόκο, την Τουρκία. Δεν θα πρέπει αυτό που συμβαίνει με την Νότια Αφρική να συμβεί και με άλλες περιοχές ε, και με άλλε τρίτε χώρε. Θα πρέπει να σεβαστούμε του καταναλωτέ μα, αλλά και του παραγωγού μα, του γεωργού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Δεν ζήτησε άλλο κανεί το λόγο, οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Ζωάν Ονοφρέ, για να απαντήσει. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από στην Αντιπρόεδρο Αγγίλερα εάν παρεξηγήθηκε η πρώτη μου παρέμβαση και θεωρήθηκε ότι είναι ισπανική η κρίση και το πρόβλημα. Συμφωνώ. Είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα και η κρίση και εμείς η Κομισιόν έχει καταστήσει σαφές ότι η κατάσταση Το τομέα των εσπεριδοειδών είναι δραματική. Έχουμε αναφέρει τους λόγους ε, για τους οποίους οι τιμές είναι χαμηλές. Δεν είναι τόσο χαμηλές όσο λένε οι ευρωβουλευτές. Οι ισπανικές αρχές μας λένε πολύ υψηλότερες ε, τιμές από ό,τι ακούστηκε εδώ. Οπότε ε, καλό είναι να τις ελέγξετε. Επίσης ήμουν σαφής ε, και είπα τους αριθμούς σε σχέση με τις νότιο-αφρικανικές εισαγωγές. Οι λόγοι της κρίσης ε, δεν οφείλονται στις εισαγωγές από την Αφρική. Όχι, είτε μας αρέσει είτε όχι. Οι αριθμοί δεν δείχνουν σημαντική αύξηση των εισαγωγών πορτοκαλιών από την Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια της περίοδου που είναι κρίσιμη για την ευρωπαϊκή παραγωγή. Έχουμε ακριβώς διαπραγματευτεί αυτή τη συμφωνία για να μην συμπίπτει με την ευρωπαϊκή παραγωγή. Και σε σχέση με την υποτιθέμενη στρέβλωση του ανταγωνισμού από το γεγονός ότι οι νοτιοαφρικανοί παραγωγοί χρησιμοποιούν διαφορετικά οκτώνα, Θα αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπε ο Επίτροπος ε, Χόγκαν εδώ ότι στις εμπορικές μας συμφωνίες δεν διαπραγματευόμαστε χαμηλότερες ποιοτικές προδιαγραφές. Πρέπει όλες οι αγωγές να σέβονται τις φυτοϊγειονομικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Αγγιλέρα. Ελπίζω να κρατήσω ακόμη για λίγο τη φωνή μου. Μπορεί να μου πει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί πέραν των συγκεκριμένων στοιχείων για τι αγωγές σε ένα συγκεκριμένο μήνα, αυτό που προβληματίζει τους γεωργού μας είναι το θέμα της αμοιβαιότητα. Δηλαδή, ο έλεγχο που γίνεται στα τελωνία. Μου είπε σήμερα το πρωί ένα γεωργό, με ρώτησε μάλλον, πώς είναι δυνατόν εμείς να πουλάμε πορτοκάλια στι Ηνωμένε Πολιτείε και να έχουμε μόνο δύο λιμάνια εισόδου για να διαθέσουμε τα προϊόντα μα στι ΗΠΑ. Μόνο δύο λιμάνια εισόδου υπάρχουν στι ΗΠΑ. Ενώ για την εισαγωγή πορτοκαλιών από την Νότια Αφρική, ε, από την Αίγυπτο, από την Τουρκία ή από οπουδήποτε αλλού, έχουμε 100-150 λιμένες εισόδου. Δεν ξέρω πόσα λιμάνια έχουμε στην Ευρώπη. Όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια είναι λιμάνια εισαγωγής για εισαγόμενα προϊόντα. Οπότε είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα. Μπορεί να έχουμε κάποιους γενικούς κανόνες, αλλά η τελωνιακή έλεγχη δεν είναι ίδια σε όλα τα λιμάνια. Και η είσοδος επίσης ε, είναι άνηση, λόγω των άνησων απαιτήσεων που εφαρμόζονται. Υπάρχουν προβλήματα λοιπόν. Με το λιμάνι του Ρότερνταμ. Υπάρχουν προβλήματα στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Το έχω καταγγείλει και στο παρελθόν. Και το επαναλαμβάνω. Πώς είναι δυνατόν για να πουλήσουμε ε, στις ε, Ηνωμένε Πολιτείε, ε, οτιδήποτε, ντομάτες, αγκούρια, πορτοκάλια, όλα τα εισαγόμενα προϊόντα εισέρχονται από δύο μόνο λιμάνια και έτσι διευκολύνονται οι έλεγχοι, ενώ εμείς έχουμε ένα σωρό. Μπορεί να μου πει εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν οι κοινωνικέ περιβαλλοντικέ απαιτήσει Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντίστοιχε με αυτέ τη Νοτιοαφρική, γιατί από ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον δεν είναι ίδιε οι απαιτήσει τη Νοτιοαφρική με τι δικέ μα. Έχουμε προϊόντα που απαγορεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλα αυτά επιτρέπονται στην Νότια Αφρική. Στην Αίγυπτο, στην Νότια Αφρική επιτρέπονται ουσίες που εμείς έχουμε απαγορεύσει και προϊόντα που εμείς έχουμε απαγορεύσει. Οπότε ουσιαστικά εισέρχονται απαγορευμένα προϊόντα ή προϊόντα με απαγορευμένες ουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ισχύουν λοιπόν όλοι οι, κανόνες, οι ίδιοι κανόνε για όλου. Εξού και η ανισότητα, η άνηση μεταχείριση. Οι παραγωγές περιδοειδέν δεν, έχουν, δεν φοβούνται τον ανταγωνισμό. Αλλά θέλουν θεμητό ανταγωνισμό, με ισότιμου όρου ανταγωνισμού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνε παραγωγή και από τη στιγμή που δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνε παραγωγή, η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη και άδικη. Και δεν ισχύει αυτό μόνο με τα εσπεριδοειδή. Το πρόβλημα είναι ότι ο έλεγχος στα τελωνία είναι ανεπαρκής. Υπάρχουν διαφορετικές επίσης διατάξεις εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολλά θέματα, εξού και διαφοροποιημένη δυσμενής μεταχείριση προς τους Ευρωπαίους γεωργούς. Και αυτό σας ρωτάω λοιπόν. Μπορείτε να μου εγγυηθείτε ότι οι περιβαλλοντικές διατάξεις και οι διατάξεις περί στην Νότια Αφρική είναι αντίστοιχες ή παρόμοιες με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να μου το εγγυηθείτε. Από ό,τι ξέρω δεν ισχύουν οι ίδιες διατάξεις και οι ίδιες προδιαγραφές. Και επίση, η πρόσβαση μέσω των λιμένων, ε, η εθνική έλεγχη, η εθνική τελωνιακή έλεγχη είναι διαφορετική και η εφαρμογή των ε, κανόνων είναι διαφορετική. Άλλε τρίτε χώρε έχουν ένα-δυο λιμάνια μόνο για τι εισαγωγέ του. Εμεί έχουμε 100 και λιμάνια. Εκεί θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση στου τελωνιακού ελέγχου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είναι σαν να γίνεται διάλογος κουφών για αυτό το θέμα. Γιατί αν δεν αναλύουμε τον κόσμο και τα στοιχεία που έχουμε με τον ίδιο τρόπο για να το ξεπεράσουμε αυτό είναι να σας καλέσουμε στην ε, Βαλένσια για να διαπιστώσετε ακριβώς τι συμβαίνει. Να έρχεται σε επαφή με την κυβέρνηση της ε, Βαλένσια και με τις οργανώσεις των Γεωργών για να μάθετε από πρώτο χέρι τι συμβαίνει. Ε, και να δούμε ποια είναι τα αίτια, αν είναι τα, αυτά που λέμε εμείς ή αυτά είναι αυτά που είπατε εσείς αποκλειστικά. Επί τόπου διαφορετικά ε, θα καταλάβουμε όλοι μαζί ακριβώς τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Μάλιστα, εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πάλι. Πολύ ευχαρίστω θα έρθω στη Βαλένθια, αφόσον με καλείτε. Ε, Για το συγκεκριμένο θέμα της Αντιπροέδρου, κύριε Αγγιλέρα, υπάρχουν δύο ζητήματα που θα ήθελα να τονίσω. Το πρώτο είναι πράγματι έχουμε μια εμπορική συμφωνία με κάποιες, κάποιες ε, τρίτες χώρες, αναφέρατε τις ΣΥΠΑ. Δεν έχουμε εμπορική συμφωνία με τις ΣΥΠΑ. Οπότε ε, λογικό είναι να έχουμε διαφορετικές συνθήκες πρόσβασης και επιβεβαιώνω επίσης ότι οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες δεν είναι οι ίδιες με αυτές που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο έχει σημασία εδώ σε σχέση με τις εμπορικές συμφωνίες δεν είναι αυτό, είναι το ότι οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κανόνες ε, για κατάλοιπα ζυζανιοκτώνων πρέπει να σέβονται ακριβώς τις ίδιες συνθήκες με τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Αυτό είναι το θέμα. Και τέλος, θα ήθελα να τονίσω και πάλι, ανεξαρτήτως ε, του, δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία αυξημένων εισαγωγών πορτοκαλιών από την Νότια Αφρική στην περίοδο η οποία βλάπτει την παραγωγή σας. Σας ευχαριστούμε. Είναι πολύ φλέγον αυτό το θέμα και επίκαιρο της, τη σύναψη των εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, δεν θα πρέπει να εισάγουμε προϊόντα που διαταράσσουν ή στρεβλώνουν την ενιαία αγορά. Σήμερα έχουμε αυτό το πρόβλημα με τα σπεριδοειδή που δεν είναι ισπανικό αλλά πανευρωπαϊκό. Η εμπορική συμφωνία θα πρέπει να είναι αμοιβαία επωφέλης για όλα τα συμβαλόμενα μέρη, όχι μόνο για τη μία πλευρά και ταυτόχρονα μπορεί να μας ευνοεί οικονομικά η μια εμπορική συμφωνία, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να προστατεύουμε και την ακαιρεότητα τη ενιαίας μας αγοράς. Μην το ξεχνούμε. Κυρία Αγγιλέρα, πολύ σύντομα παρακαλώ. Μάλιστα, μόνο επειδή ολοκληρώνω τη συζήτηση να πω ότι φαίνεται και ακούγεται σαν διάλογο σκουφών, αλλά εγώ θέλω να τονίσω ότι είναι παρόντε σε αυτή τη συζήτηση εκτό από του εκπροσώπου ε, του τομέα, η σύμβουλο ε, τη Περιφερειακή Κυβέρνηση τη Βαλένσια και η, αντι... Ε, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου που εργάζονται μαζί σε συνεργασία με όλων των τους εκπροσώπους του, του τομέα έχουν έρθει μια-δύο φορές εδώ ε, χέρι-χέρι με τους εκπροσώπους ε, του τομέα των εσπεριδοειδών για να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα, τα προβλήματα. Κάνει πολύ σπουδαία δουλειά η περιφερειακή κυβέρνηση σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση της χώρας για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ ολοκληρώνω αυτό το σημείο, θα ήθελα να παρακαλέσω, αν γίνεται, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έρθει σε επαφή και με Γιώργους και εκπροσώπους του κλάδου αυτού που βρίσκονται και στην αίθουσα για να διαμορφώσει καλύτερη γνώμη. Θα θέλαμε ιδιαίτερως να συνεχιστούν οι συζητήσεις μεταξύ σας με τους εκπροσώπους του κλάδου, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Έχουμε τώρα μια άλλη σημαντική ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Διευθυντή Κλάρκ για τα, τις εμπορικές συμφωνίες και τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργούν στην Γεωργία. Βέβαια, το διεθνές εμπόριο και σχετικές διαπραγματεύσεις είναι καθήλια αρμοδιότητα της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Ε, επηρεάζουν όμως και γεωργικά προϊόντα και μάλιστα κάποια ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα. Γι' αυτό και ενδιαφερόμαστε και εμείς για τις ε, εμπορικές συμφωνίε. Υπάρχει μια διαμάχη σύγκρουση αρμοδιοτήτων πολλές φορές με την Επιτροπή ΙΝΤΑ για τα θέματα αυτά, γιατί θα πρέπει και η φωνή των γεωργών να ακούγεται για θέματα που επηρεάζουν την ε, αγορά. Γι' αυτό και καλέσαμε τον Διευθυντή, τον κύριο Τζον Κλάρκ, για να μας ενημερώσει για διάφορες εμπορικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή και πώς επηρεάζουν την κοινή μας αγορά. Γιατί η κοινή αγορά είναι τεράστια αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει όμως να την προστατεύσουμε. Έχουμε επιγνωσεί ότι η εμπορική συμφωνία δεσμεύει όλα τα συμβαλόμενα μέρη, αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις μας. Θα ήθελα λοιπόν κύριε Κλάρκ, να μιλήσουμε και για το τι που έχει βέβαια ανασταλεί, αλλά ανεπίσημα ακούμε ότι γίνονται διάφορες διαπραγματεύσεις που εμπλέκουν και το γεωργικό τομέα. Πώς έχουν λοιπόν οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Επίσης, θα ήθελα να μας μιλήσετε για την επαναφορά των τελωνιακών δασμών για το ρύζι. Μας ενημέρωσε η Επίτροπος Μάνστρομ στην Ολομέλη για το θέμα αυτό για τα προϊόντα, για το ρύζι από την Καμπότζη και τη Μιαμάρ. Επίσης, τι γίνεται ε, στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για για την περίφημη, το περίφημο παραθυράκι που υπήρχε για τον τρόπο που γινόταν ο τεμαχισμός των ε, ε, πουλερικών, ώστε να ακόμη και ευγενή κομμάτια κρέατος πουλερικών να ε, με τη διαφορετική κοπή να εμπίπτουν σε χαμηλότερη δασμολογική κατηγορία και άρα να δημιουργούν πρόβλημα στην αγορά με τις χαμηλότερες τιμές. Ελπίζω να καταφέραμε να κλείσουμε αυτό το ατυχές παραθυράκι που χρησιμοποιήθηκε εκτενώς. Επίσης, ε, Ε, από την Ουκρανία. Κυρίως ε, προϊόντα τέτοια φτάνουν στις κοντινές χώρες, πρώτα απ' όλα στην ε, Πολωνία, αλλά μετά κυκλοφορούν και στις υπόλοιπε περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε νέα αγορά, οπότε τα, τα προϊόντα κυκλοφορούν ελεύθερα. Άρα θα μας ενδιαφέρει η σε ελεύθερων συναλλαγών με το Mercosur και για τα θέματα του βοήου ενδιαφερόμαστε εκεί και πολυερικών επίσης. Επίσης, τι γίνεται με τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Και τέλος, πείτε μας δύο λόγια και για το Brexit. Πολύ ευαίσθητο αυτό το θέμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν θα θέλαμε να βγούμε χαμένοι ούτε εμείς ούτε η Μεγάλη Βρετανία και φυσικά ούτε η Βόρεια Ιρλανδία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Κύριε Κλάρκ, περιμένουμε τις πληροφορίες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την τελευταία φορά που ήρθα είχαμε αρκετές εξελίξεις στο μέτωπο του εμπορίου Πρώτα απ' όλα έχουμε τέσσερις εμπορικές ε, συμφωνίες ε, που έχουν ουσιαστικά συναυθεί και προσεχώς θα τεθούν ενισχύ. Ε, με την Ιαπωνία, 1η Φεβρουαρίου, με την Σιγκαπούρη που ψηφίζεται από την Επιτροπή Ίντα σήμερα, η συμφωνία με το Βιετνάμ που ολοκληρώνεται θα τεθεί ενισχύ μέχρι το τέλος του έτους και με το Μεξικό επίσης ε, πριν το τέλος ε, του έτους. Όλες αυτές οι συμφωνίες, η Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Βιετνάμ, Μεξικό, είναι καλοδεχούμενες από τα κράτη-μέλη μας και από τους ενδιαφερόμενους, την Συνομοσπονδία των Αγροτών και τις ε, Γεωργικές Ενώσεις και παρέχουν πολλά ωφέλη για τους εξαγωγείς τροφίμων, προστατεύουν και τις 200-300 γεωγραφικές ενδείξεις ε, σε όλες αυτές τις αγορές, οπότε πρέπει να τις βλέπουμε θετικά, ειδικά την Ιαπωνία, που είναι το 30% του παγκοσμίου εμπορίου Ευρωπαϊκή Ένωση Ιαπωνία, η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία ε, πέρα από την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για τους ε, γεωργούς μας όσον αφορά τις συνεχιζόμενες εμπορικές διαπραγματεύσεις ε, με το Mercosur. Η πρόοδος εκεί είναι περιορισμένη, θα χαρείτε ίσως. Δεν ξέρουμε πότε θα συνεχθεί η συμφωνία. Δεν ξέρω εάν υπάρχει το κατάλληλο πολιτικό κλίμα για να καταλήξουμε σε μια τέτοια συμφωνία και εν των ευρωεκλογών. Οπότε δεν το βλέπω προσεχώς. Υπάρχει και η νέα βραζιλιανική κυβέρνηση που δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει την θέση της ε, για το θέμα αυτό. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των θέσεων των δύο πλευρών ε, για την γεωργία. Πρέπει να έχουμε κάποια σοβαρή προσφορά από το Μερκοσούρ για τις δικές μας προτεραιότητες, κρασί, γαλακτοκομικά, ελαιόλαδο, πριν σημειωθεί κάποια πρόοδος. Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία τα αναφέρατε, είναι νωρίς ακόμα, δεν έχουμε καν ανταλλαξή κάποιες πρώτες προσφορές πρόσβασης στις αγορές, οπότε νομίζω ότι θα περιμένουμε για μετά το καλοκαίρι. θα συζητήσουμε πρόσβαση στην αγορά μόνο εάν δούμε κάποια πρόοδο από τη δικιά τους την πλευρά μετά. Στην Ασία επίσης ε, οι διαπραγματεύσεις με την Ινδονησία είναι κάπου στη μέση θα έλεγα αλλά επιβραδύνονται λόγω της ευρωπαϊκής θέσης ε, για το φινικέλαιο και την αποδάσωση που ενοχλεί τους Ινδονησίους Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη έχουν ε, ανασταλεί διαπραγματεύσεις για λόγους ανθρωπινών δικαιωμάτων και η Μαλαισία σταμάτησαν αυτή τις διαπραγματεύσεις γιατί δεν θεωρούν ότι είναι προς το συμφέρον τους. Νομίζω ότι θα αλλάξουν άποψη όταν τεθεί ενισχύ η συμφωνία με το Βιετνάμ και θα έχει πλέον το Βιετνάμ ένα πλεονέκτημα. Η ΕΠΑ, αναφέρατε τη ΕΠΑ κύριε Πρόεδρε, παρουσιάσαμε στο Συμβούλιο μια διαπραγματευτική έντολη για την συμφωνία με τις παλαμόνο μόνο για βιομηχανικούς δασμούς, τίποτα για τα μη δασμολογικά εμπόδια και τίποτα για την γεωργία. Αυτό νομίζω αντικατοπτρίζει την συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Γιούνκερ το καλοκαίρι για να δούμε πώς θα διαπραγματευτούμε μια περιορισμένη συμφωνία η οποία θα καλύπτει μόνο τα βιομηχανικά προϊόντα και τους δασμούς. Σαφώς αποκλείεται η γεωργία, όπως ήταν και από την πλευρά των ΙΠΑ, για τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις ε, ναυτιλιακές υπηρεσίες. Έχουμε λοιπόν μία εντολή την οποία ελπίζουμε να εγκρίνει το Συμβούλιο. Οι ΙΠΑ επίσης ε, οριστικοποιούν ε, την δική τους διαπραγματευτική εντολή που είναι τελείως διαφορετική από τη δική μας Εκεί πέρα δίνεται προτεραιότητα στη γεωργία, δίνεται προτεραιότητα στον κανονισμό SPS. Ουσιαστικά είναι μια δεύτερη TTIP και ειλικρινά είναι δύσκολο να δούμε πώς θα συμβιβάσουμε δύο διαμετρικά αντίθετες στάσεις και ε, εάν ε, επιβληθούν ε, δασμοί στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και ανταλλακτικά τον Μάρτιο θα δηλητηριάσει τελείως το κλίμα, κάτι τέτοιο, ακόμα και για τα βιομηχανικά αγαθά. Αναφέρατε κάποια άλλα θέματα, διμερή κύριε Πρόεδρε, η Ουκρανία, έχουμε μία εντολή διαπραγμάτευσης για τις μελλοντικές εξαγωγές πουλερικών θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα και σκοπεύουμε να επιβληθεί ένα πλαφόν στις εξαγωγές ε, στήθους ε, πουλερικών ε, και έτσι να μπει και αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι του ζώου εντός των δασμών. Προσεχώς νομίζω. Και θα κλείσει αυτό το παραθυράκι. Για τη είπα και πάλι διαπραγματευόμαστε μια συμφωνία με τη ΣΥΠΑ για το κρέας χωρίς ορμόνες και την σχετική ποσόστοση για να πάει ένα κομμάτι της ποσόστοσης μόνο στη ΣΥΠΑ. Οι συζητήσεις μας είναι σε προχωρημένο στάδιο και ελπίζω να καταλήξουμε σε κάποιες εβδομάδες και όχι μήνες. Εάν δεν επιτύχουμε συμφωνία με τις ΗΠΑ, τότε ξαναπάμε στις κυρώσεις επί των ευρωπαϊκών εξαγωγών και την ακύρωση της ποσόστοσης ολόκληρης. Είναι τόσο απλό. Ο τομέας του ρυζιού. Οι εξαγωγές της Καμπότζης και της Μιανμάρ. Αυτό το συζητήσαμε 18 Ιανουαρίου, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, και η αδασμολόγητη πρόσβαση του ρησιού αντικαθίσταται από έναν δασμό 175 ευρώ στον τόνο, που σε τρία χρόνια θα έχει πέσει στα 125 και θα εκπνεύσει. Η δράση αυτή είναι δικαιολογημένη Σπανιότατα η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κάτι τέτοιο, αλλά στην περίπτωση αυτή είναι δικαιολογημένη. Η τιμή ή μάλλον το ποσοστό της αγοράς ε, του ρυζιού των Ευρωπαίων παραγωγών έχει μειωθεί στο μισό από το 60% στο 30% τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ ταυτόχρονα οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 90%. Ε, υπήρχε μια σαφής ε, αιτιώδης ε, σχέση μεταξύ των φθηνών εισαγωγών από αυτές τις δύο χώρες και του χαμηλού ποσοστού της αγοράς των Ευρωπαίων παραγωγών. Οπότε ακολουθήσαμε το γράμμα και το πνεύμα της συμφωνίας τα πάντα πληνόπλων για να υπάρξει αυτό το μέτρο για δύο χρόνια. Τέλος, μια διμερής ε, περίπτωση, οι ισπανικές επιτραπέζιες ελιές, ξέρετε πως οι ΙΠΑ έχουν επιβάλει μια τελείως αδικαιολόγητη θεωρούμε εμείς ε, και παράνομη κύρωση, έναν δασμό κατά των επιδοτήσεων για τις επιτραπέζιες ελιές ε, της Ισπανίας και ετοιμάζουμε μια προσφυγή στον ΠΟΕ κατά τον ΙΠΑ για να φύγει αυτός ο δασμός. Κάποια πράγματα ακόμα. Ο ΠΟΕ Εργαζόμαστε εκεί σε τρία μέτωπα. Πρώτα απ' όλα να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα επίλυσης διαφορών, να εισαχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια. Δεύτερον, μαζί με τις ΙΠΑ, Ιαπωνία και λοιπούς, να αναπτύξουμε ισχυρότερους κανόνες για τις βιομηχανικές επιδοτήσεις, την υποχρεωτική μεταφορά τεχνολογίας και την κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας ε, και τρίτον υπάρχουν διαπραγματεύσεις που γίνονται για την αλληλεία, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την γεωργία. Δεν αναμένω στον ΠΟΕ κάποιες ε, διαπραγματεύσεις ε, που θα λάβουν χώρα για το επόμενο έτος. Πιθανώς μετά την επόμενη Υπουργική Διάσκεψη στα μέσα του 2020 οι στόχοι μας παραμένουν οι ίδιοι να αναπτύξουμε ισχυρότερους κανόνες για να μειώσουν όλα τα μέλη του ΠΟΕ τις στηρίξεις που διαστρεβλώνουν το εμπόριο, ενώ να παραμείνει ανέπαφο το πράσινο κουτί οι άμεσες πληρωμές δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το Brexit κύριε Πρόεδρε, διστάζω λίγο να μπω στο θέμα αυτό. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνήσει, το οποίο δεν είναι καθόλου σίγουρο στην συμφωνία αυτή, τότε θα έχουμε επιγής ειρήνη ας πούμε για κάποια χρόνια και ελπίζουμε το εμπόριο γεωργικών και τροφίμων ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο να μην διαταραχθεί. Ε, θα παραμείνει ουσιαστικά στην ενιαία αγορά και την τελωνιακή ένωση στο ΕΒ μέχρι να προκύψει μια νέα συμφωνία ό,τι μορφή και αν έχει. Εάν πάμε σε Brexit χωρίς συμφωνία στις 29 Μαρτίου τότε θα, οπωσδήποτε θα υπάρχει μια διατραχή τεράστια στον κλάδο. Οι 27 εξάγουν 40 δισεκατομμύρια ευρώ ε, τέτοιων προϊόντων στο ΕΒ Το Ηνωμένο εξάγει 15 δισεκατομμύρια ευρώ το έτος ε, στην ε, Ήπειρο στους 27. Μεγάλος όγκος εμπορίου, ειδικά για ζωικά προϊόντα, τα οποία έχουν αρκετά ψηλούς δασμούς σε κάποιες περιπτώσεις και βεβαίως σοβαρούς υγειονομικούς ελέγχους. Στην περίπτωση λοιπόν ενός Brexit χωρίς ε, συμφωνία ε, ίσως ε, εισαχθούν δασμοί νομικά θα είναι αναπόφευκτο για να επιβάλλουμε τις υποχρεώσεις μας ε, σύμφωνα με τον ΠΟΕ και εμείς και το Ηνωμένο Βασίλειο και θα υπάρχουν έλεγχοι υγειονομικοί επιθεωρήσεις των φορτίων για να είμαστε σίγουροι ότι συμμορφώνονται και πιθανώ το, το Ηνωμένο Βασίλειο θα κάνει το ίδιο στα δικά του λιμάνια. Οπότε το κόστος θα είναι τεράστιο και η διατάραξη του εμπορίου. Ε, επεξεργαζόμαστε όλα αυτά τα σενάρια στην Κομισιόν για να είμαστε έτοιμοι. Εντό ε, της ε, ΚΑΠ έχουμε κάποια μέσα, κάποια εργαλεία. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε ο εκπρόσωπο εδώ πέρα τη Κομισιόν. Στην διάθεσή μας λοιπόν για να περιορίσουμε τον αντίκτυπο όπως έγινε παραδείγματος μετά το ρωσικό εμπάργκο στις ευρωπαϊκές εξαγωγές ύψους 6 δισεκατομμυρίων. Πέρα από αυτό ο αντίκτυπος στους παραγωγούς θα είναι πολύ σοβαρός. Σας ευχαριστούμε κύριε Δευθυντά. Θα ακολουθεί η συζήτηση, όπως είπαμε. Πρώτο, ο κύριος Χόισλινγκ. Äh, σας ευχαριστώ κύριε Κλάρκ ε, που ήρθατε. Ε, παρακολουθήσατε και την προηγούμενη συζήτηση και ε, μας είπε ο εκπρόσωπος σας το πρωί ότι δεν υπάρχει dumping μέσω των εισαγωγών από τις συμφωνίες ελευθερου εμπορίου. Γεγονός είναι ότι υπάρχει, αλλά Τώρα για την ε, TTP παριθμών 2. Θεωρώ ότι όπως είπατε και εσείς ε, άλλωστε ε, μπορούμε να έχουμε διάφορα προβλήματα με τις Εντάξει αυτά είναι προβλέψιμα βεβαίως Δεν νομίζω πάντως είπα να πούν τελικά θα αφήσουμε τον ε, γεωργικό τομέα εκτός. Επενέσατε συγκεκριμένα την Ιαπωνία πράγματι. Βεβαίως η Ιαπωνία κατάφερε αμέσως να ξαναρχίσει την ε, εμπορική αλληλεία φαλενών. Για το Βιετνάμ υπάρχει η υποψία, η αιτιολογημένη υποψία ότι η συμφωνία αυτή με το Βιετνάμ σημαίνει ότι υπάρχει ξύλο προϊόν λάθρο υλοτομίας το οποίο αλλάζει η ετικέτα προέλευσης και μετά εξάγεται ως βιετναμέζικο. Πρέπει να εμποδιστεί αυτό. Αυτό το οποίο πραγματικά με ενοχλεί και με εκνευρίζει ε, είναι η υπόθεση με το Μερκοσούρ και λέτε ότι δεν θα προχωρήσει λόγω ευρωεκλογών. Ε, συγγνώμη, λόγω των ευρωεκλογών είναι σκανδαλώδες ε, το ότι ε, συνεχίζουμε να διαπραγματευόμαστε με τον ακραίο δεξιό Μπολσονάρου ή τι το αγνοούμε απλώς να πούμε α ναι συγγνώμη εμείς έχουμε μια εντολή και συνεχίζουμε τη διαπραγμάτευση. Είπατε αντιθέτως ότι διακόψαμε τις συνομιλίες με άλλες χώρες λόγω ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ με τον Μπολσονάρο δεν συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή απορώ. Δύο φορές ε, έχει απευθύνει ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, επιστολή, ο Μογκερίνη, μάλλον εμείς απευθύναμε επιστολή, ε, πως θα έπρεπε κάποια στιγμή να δείξουμε ότι δεν μπορεί να παριστάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Για τις εισαγωγές βοηδών και τα σχετικά, αν δεν υπάρξει κάποια πολιτική αλλαγή. Δεν μπορώ να παριστάνω ότι δεν έχει υπάρξει μια πολιτική αλλαγή όμως. Πραγματικά δηλαδή δεν, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Έχετε να μας πείτε κάτι. Ευχαριστώ κύριε Ντελαέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ λακωνική. Θα σας πω κάτι απλούστατο. Ας μην εισάγουμε ε, τη γεωργία και το τρόφιμα που στην Ευρώπη ε, δεν δεχόμαστε. Κάτι που δεν θέλουμε στην Ευρώπη είναι κρίμα να το εισάγουμε έξωθεν. Επίσης, ε, με το θέμα του βιοντίζελ από την Αργεντινή τι γίνεται. Κύριε Αγγιλέρα, ευχαριστώ. Και καλώς ήρθατε κύριε Κλάρκ. Ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα κατατόπιση που μας κάνατε και την πορεία των διαπραγματεύσεων. Μόλις πριν από λίγο μιλήσαμε για τον αντίκτυπο που έχουν οι εισαγωγές ε, εσπεριδοειδών, κυρίως από την Νότια Αφρική, στον κλάδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη ε, πειράζουν πολύ αρνητικά τον κλάδο εισαγωγές από την Νότια Αφρική και στο μέλλον φοβούμαστε ότι θα τον ε, πλήξουν ακόμη περισσότερο. Το πρόβλημα που έχουμε με τις εμπορικές συμφωνίες όλο και περισσότερο έγινε στη διαφορά στι απαιτήσει που έχουμε από την ευρωπαϊκή παραγωγή και από τις ε, παραγωγές των τρίτων χωρών. Γιατί αν όντω εφαρμοστεί ε, η αμοιβαιότητα και οι ίδιες προδιαγραφές και απαιτήσει που ισχύουν στην Ευρώπη για την παραγωγή εσπεριδοειδών ή ε, οποιοδήποτε άλλο προϊόντος, θα πρέπει να είναι αντίστοιχε και στις τρίτες χώρες είναι διαφορετικέ και οι κλιματικέ συνθήκε, αλλά και οι απαιτήσει και οι προδιαγραφέ στι τρίτε χώρε. Εμεί είμαστε μια πολύ απαιτητική κοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε πολύ υψηλέ φυτοϊγειονομικέ απαιτήσει και προδιαγραφέ και πολύ καλά κάνουμε. Αλλά αντίστοιχο θα πρέπει να απαιτούμε και από τι τρίτε χώρε που, εισάγουν που εξάγουν προϊόντα προ εμά. Γιατί διαφορετικά δημιουργείται μία άνηση μεταχείριση και μία δυσμενή μεταχείριση και ένα dumping ει βάρο των δικών μα παραγωγών. Ε, είναι πολύ ευπρόσδεκτο το μέτρο που λάβατε για την επαναφορά των δασμών για το ρύζι. Αλλά δυστυχώς ε, δεν ε, αξιολογήθηκε δεόντως την στιγμή που έπρεπε οι επιπτώσεις αυτών των εμπορικών συμφωνιών με τις χώρες της Δυτικής Ασίας στο ρύζι. Και αυτό πληρώνουμε τώρα. και έφτασε ο κόμπος το χτένι με τους ε, οριζοπαραγωγούς να υφίστανται τα πάνδυνα λόγω των μαζικών εισαγωγών. Ε, βέβαια, μερικά πράγματα εκφεύγουν τι δικέ αρμοδιότητε, αλλά επιμένω στην απέτηση τη αμοιβαιότητα. Έχουμε κάποιου κανόνε θα πρέπει να πετούμε να εφαρμόζονται και στους, από του εταίρου μα. Επίση, η τελωνιακή έλεγχη. Η, τα τελωνία είναι εθνική αρμοδιότητα και κάθε κυβέρνηση διαφορετικά εφαρμόζει την κοινοτική νομοθεσία. Επιπλέον, τα κράτη-μέλη και, και οι περιφέρειες διαπραγματεύονται επιμέρου επιμέρους πρωτόκολλα. Πέρα των συμφωνιών μπορούν να διαπραγματεύονται και πρωτόκολλα στα οποία ισχύουν διαφορετικοί κανόνε. Με τι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουμε συμφωνία. Μακάρι να μην συνάψουμε καμία συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ και να κρατήσουμε τι αποστάσει μα. Αλλά στι Ηνωμένε Πολιτείε έχουμε μόνο δύο λιμάνια εισόδου για τα πορτοκάλια. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισαγόμενα πορτοκάλια από οποιαδήποτε χώρα, έχει 150 λιμάνια να διαλέξει την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπει στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Είναι θέμα λοιπόν ε, συμφωνιών, επιμέρους πρωτοκόλων και τελωνιακών ελέγχων που είναι διαφορετικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που επιβαρύνουν μαζί με την έλλειψη της αμοιβαιότητας τους γεωργούς μας. Ευχαριστώ κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ κύριε Κλάρκ που ήρθατε. Πραγματικά είναι καταθλιπτικό το πόσοι σας παρακολουθούν δεδομένης της ε, αρχαιότητάς σας και του βαθμού σας. Χαίρομαι που ακούω ότι η Κομισιόν παίρνει στα σοβαρά πλέον την προοπτική ενός Brexit χωρίς ε, συμφωνία ή με τους όρους του ΠΟΕ. Μας δώσατε τους αριθμούς. Έχουμε ένα κενό 25 εκατομμυρίων, ε, δισεκατομμυρίων ευρώ σε τρόφιμα. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των όσων πουλάει και εισάγει η Μεγάλη Βρετανία. Τα 25 αυτά δισεκατομμύρια είναι πολλές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζω ότι ε, όσοι βλέπουν τις δουλειές τους να κινδυνεύουν θα αρχίσουν να ασκούν πίεση στους κυρίους Γιούνκερ και Μπαρνιέ για να μην υπάρξει ε, χάος και η πολιτική να περάσει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με πιο ρεαλιστικά ζητήματα όπως το βιός των Ευρωπαίων αγροτών. Ε, τώρα ακούγονται διάφορα τρομοκρατικά πράγματα στη Βρετανία. Μιλάνε για έλλειψη τροφίμων ε, και φαρμάκων. Θα γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τους ε, κανόνες του ΠΟΕ και με άλλες χώρες. Και αν αντιλαμβάνομαι σωστά δεν εξάγεται φάρμακα σε αυτές τις χώρες ή τρόφιμα. Η τι γίνεται, είναι τόσο δύσκολο που δεν ε, μπορεί να γίνει τίποτα. Αλλά εμείς εξάγουμε φάρμακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, φάρμακα χρειάζονται όλοι και συνήθως γρήγορα. Και ελπίζω, τουλάχιστον ω προς αυτό, να υπάρξουν κάποιες γρήγορε αμοιβαίε διευθετήσει τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ. Κύριε Σουλαζό. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας πω μόνο πως μάθατε πως η Ευρωπαϊκή ε, Γεωργία αποκλείεται από κάθε εμπορική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Επιτέλους, όμως αντίθετα οι εισαγωγές αυξήθηκαν, αυξήθηκαν 112% το τελευταίο εξάμεινο από τη ΣΥΠΑ. Μάλιστα και άλλες αυξήσεις που προβλέπονται προσεχώς. Μεγάλη δε εξάρτηση έχουμε από την Αμερική. Αυτό είναι αντίθετο με το στόχο της κοινή γεωργική πολιτικής, δηλαδή ε, τροφική αυτονομία και ε, κυριαρχία. Χωρίς να μιλήσουμε βέβαια για την περιβαλλοντική πολιτική τον είπα, ενώ η Κομισιόν θέλει να επιβάλλει ακόμη περισσότερους κανόνες ε, για το περιβάλλον μέσω μιας τιμωρητικής οικολογικής πολιτικής. Γιατί λοιπόν ε, να μην αποκλείεται κάθε φορά και συστηματικά η γεωργία μας από τέτοιου είδους συμφωνίες. Πώς εξηγείται το γεγονός ε, διαρκούς επιβολής ε, επί των γεωργών μας κανόνων που δεν απαιτείται από τις τρίτες χώρες που εξάγουν προς εμάς προϊόντα που αλλιώς τα απαγορεύονταν από τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Σας ευχαριστώ. Ήρθε η ώρα σας κύριε Διευθυντά. Thank you very much. I'll, I'll try to reply to all. ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Είπα, πρώτα απ' όλα, είναι πρόθεση της ε, Κομισιόν να εξαιρεθεί η Γεωργία από οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση με τις Είπα, Αυτό το είχαμε συμφωνήσει ρητός ε, με οι πρόεδροι Τραμπ και Γιούνκερ όταν ε, συναντήθηκαν. Οπότε η εντολή μας εξαιρεί τη Γεωργία. Εντάξει, σαφές. Για την σόγια από τις ΗΠΑ ε, την χρειαζόμαστε για ζωοτροφή το οποίο συμβαίνει είναι ότι οι εισαγωγέ από Βραζιλία και Αργεντινή έχουν αντικατασταθεί από αμερικανική σόγια που είναι 15% φτηνότερη από ό,τι ήταν πριν. Οπότε η αγορά αντιδρά φυσικά στο γεγονός ότι είχε απαγορευτεί η εξαγωγή της αμερικανικής σόγιας στην Κίνα κύριος Χόισλινγκ αναφέρθηκε στα προβλήματα της συμφωνίας με την Ιαπωνία. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα εφαρμογής της ε, συμφωνίας αυτής που θα τεθεί προσεχώς Η Γεγονός είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μικρό παράθυρο για τους Ιάπωνες εισαγωγής για να ζητήσουν άδειες εισαγωγής ευρωπαϊκού τυριού. Αλλά το γνωρίζουν αυτό και κάνουν τις αιτήσει τους ε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αναφέρατε κατόπιν το Βιετνάμ και τον κίνδυνο λαθροϊλοτομίας ε, και τα προϊόντα της ε, να έρχονται στην Ευρώπη μέσω του Βιετνάμ. Υπάρχει μια ομάδα εργασίας πολύ σοβαρή ΕΠΑ, Ένωση ε, ε Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ ε, με στόχο ακριβώς την πρόληψη της ε, λαθροϊλοτομίας, κάτι το οποίο είχε συζητηθεί σε μια επιτροπή του Κοινοβουλίου χτες μόλις. Και το συμπέρασμα ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μια πολύ καλή δουλειά όσον αφορά την συνεργασία με τον Βιετνάμ για την πρόληψη αυτής της κατάστασης. Τέλος για το Μερκοσούρ θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το ποιες θα είναι οι νέες πολιτικές της Βραζιλίας σε σχέση με το περιβάλλον, την βιωσιμότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι δουλειά του Συμβουλίου να αποφασίσει εάν θα αναστείλει τις διαπραγματεύσεις με το Μερκοσούρ εάν υπάρξει σοβαρή επιδείνωση σε κάποιους αυτούς τομείς. Κύρια ε, αγγελέρα είπατε κάτι το οποίο είχε γίνει και στην προηγούμενη συζήτηση για τα εσπεριδοειδή, e ότι οι τρίτες χώρες ε, δεν χρειάζεται να συμμορφώνονται με τις δικές μας τα ε, Απλούστατα αυτό δεν ισχύει. Με ή χωρίς συμφωνία ελευθερου οι εισαγωγέ ε, οφείλουν να πληρούν τις ίδιες προδιαγραφέ όπω τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Είναι τόσο απλό, δεν υπάρχει καμία διάκριση, υπάρχει εθνική μεταχείριση. Ένα πορτοκάλι από την Νότια Αφρική πρέπει να είναι όσο ασφαλές όσο ένα από την Βαλένσια. Τι ίδιε απαιτήσει πρέπει να πληρεί. Και είμαστε πολύ υπερήφανοι για τις απαιτήσει αυτές ε, που ισχύουν στην Ευρώπη ισχύουν και για την εγχώρια παραγωγή και για τις εισαγωγές. Θα έλεγα ότι έχουμε το καλύτερο σύστημα για τα τρόφιμα με τη μεγαλύτερη χνηλασιμότητα στον κόσμο. Τι άλλο να πω. Ναι. Η ανησυχία για το ρύζι. Ξέρετε, πριν από τέσσερα χρόνια ένα κράτος μέλος μας ζήτησε να ενεργοποιήσουμε την δικλίδα ασφαλείας για να μειωθούν οι εισαγωγές από την Καμπότζη και την Μιανμάρ. Η Κομισιόν ερεύνησε. Έκανε μια σοβαρή μελέτη για το εάν υπήρχαν οι συνθήκες για κάτι τέτοιο και το συμπέρασμα ήταν όχι οι εισαγωγέ τότε δεν ε, αυξανόταν δραματικά και οποιαδήποτε αλλαγή της ε, τιμής ε, του ευρωπαϊκού ρυζιού δεν οφειλόταν στις εισαγωγές. Αυτό κρίναμε τότε με βάση γεγονότα. Η κατάσταση τώρα διαφέρει και στην περίπτωση αυτή εφαρμόσαμε τα ίδια κριτήρια και καταλήξαμε ότι ναι, πρέπει να ενεργοποιηθεί η δικλίδα αυτή ασφαλεία. Οι εισαγωγέ επηρεάζουν άμεσα την ευρωπαϊκή παραγωγή. Εξού και κινηθήκαμε. Πρέπει να εφαρμόζουμε του κανόνε ε, με τρόπο δίκαιο. Αν χρειάζεται η δικλίδα ασφαλεία, ε, την εφαρμόζουμε. Εάν οι δυσκολίε στην ευρωπαϊκή αγορά οφείλονται σε άλλου παράγοντε. πρέπει και αυτό να το αναγνωρίσουμε και να μην αποδίδουμε τα προβλήματα αλλού. Κύριε Άγνιο, Επίσης και εσείς αναφέρετε κάποια γενικά πράγματα για τους ε, κινδύνους ε, και το τι θα σημαίνει ένα Brexit χωρίς ε, συμφωνία ειλικρινά είναι κάτι στο οποίο δεν μπορώ να σας δώσω μια αναλυτική απάντηση είναι για τους ανωτέρους μου αντιλαμβάνουμε ότι γίνονται κάποιες διευθετήσεις για την παροχή φαρμάκων προς τις δύο κατευθύνσεις, αλλά διαβάζω και εγώ τις εφημερίδες όπως και εσείς. Μετά ο κύριος Λουαζό ε, εκφράσατε κάποιες ανησυχίες για τον κίνδυνο του να περιληφθεί η γεωργία σε οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική συμφωνία της Ένωσης. Όπως ε, εξήγησα, ελπίζω σαφώς, ε, η Κομισιόν δεν προτείνει να περιληφθεί η Γεωργία, ε, προτείνει να εξαιρεθεί και είμαι απολύτως πεπισμένος ότι θα το κάνει αυτό το Συμβούλιο γιατί αυτό είναι και η συμφωνία των δύο Πρόεδρων. Για το γενικότερο ερώτημα σε αν μπορεί γενικότερα να εξαιρείται η Γεωργία, η απάντηση είναι όχι. Για διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα. πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τον ΠΟΕ και να καλύπτουμε ουσιαστικά το 90% του εμπορίου. Οπότε για πολλούς εταίρους που η γεωργία είναι μεγάλο κομμάτι, αν εξαιρέσουμε τη γεωργία πέφτουμε κάτω από το 90% και δεν ε, κολλάει στον ΠΟΕ, δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Δεύτερον, ε, για πολλού ε, εμπορικού εταίρου μα, η γεωργία είναι η πρώτη προτεραιότητα και ειλικρινά θα ήταν αδύνατον να συνάψουμε συμφωνία αν δεν κάνουμε κάποια ανοίγματα στη γεωργία. Και είτε μα αρέσει είτε όχι και το έχω πει και στο παρελθόν σε αυτήν την επιτροπή, οι συμφωνίε μα με τον υπόλοιπο κόσμο δεν αφορούν μόνο τη γεωργία, αφορούν και τα βιομηχανικά προϊόντα, τι επενδύσει, τι δημόσιε προμήθειες, τι υπηρεσίες. Έχουμε και άλλου κλάδου ε, που έχουν ένα ενδιαφέρον πρέπει να παραδεχτούμε ότι η γεωργία είναι μέρος των διαπραγματεύσεων, ειδικά όπου είναι η πρώτη προτεραιότητα των άλλων χωρών. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι έχουμε πλέον ένα ενδιαφέρον συμφέρον στο να περιληφθούν οι συμφωνίες αυτές ε, και να περιλαμβάνουν τη Γεωργία, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όλο και πιο ανταγωνιστική στι παγκόσμιε αγορέ. Δεν αναφέρομαι τώρα στι δυσκολίε τη εσωτερική αγορά με τι τιμέ, αλλά όταν μιλάμε για τι εξαγωγέ, είμαστε ο μεγαλύτερο εξαγωγέα τροφίμων γεωργικών προϊόντων. Έχουμε μεγάλο πλεόνασμα και είναι πολύ καλή η φήμη των ευρωπαϊκών τροφίμων και ποτών στις αναδυόμενες οικονομίες. Πριν από 10 χρόνια οι εξαγωγές ήταν ένα 7% της ευρωπαϊκής παραγωγής. Τώρα είναι 12,5%. Οπότε οι εξαγωγές γίνονται όλο και πιο σημαντικές ως ποσοστό της ε, συνολικής παραγωγής μας. Οπότε έχουμε κάθε συμφέρον στο να περιληφθεί η γεωργία και τα τρόφιμα τις ε, περισσότερες συμφωνίες εμπορίου για τα ποιοτικά προϊόντα, για τα γαλακτοκομικά, χοιρινά, κρασί, ελαιόλαδο, τα μεσογειακά προϊόντα και οι γεωγραφικές ενδείξεις επίσης. Ένας τρίτος λόγος για τον οποίο δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να περιλαμβάνουμε τη γεωργία. Σας ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Ολοκληρώσαμε την ημερήσια διατάξή μας. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Κλάρκ, τους βουλευτές, κύριος αυτούς που άντεξαν μέχρι τέλους. Ολοκληρώνουμε. Η επόμενη μας συνεδρία θα 29 του μηνός, ημέρα Τρίτη, στις